της Επιτροπής θα έχουμε και μία άλλη για την κατάσταση διατλαντικά όσον αφορά τις οικονομικές ρυθμίσεις. Τέλος, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη εκ των προτέρων διότι ο κύριος Τρισέ και εγώ θα πρέπει να φύγουμε ακριβώς στις 4 για να πάμε σε μια άλλη συνάντηση. Σύνεπως, τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε για να πάμε αμέσω στο σημείο 3 που είναι η δημόσια κρόαση με τον Ζαν Κλόντο Τρισέ δεν χρειάζεται καμία εισαγωγή να σας τον παρουσιάσω. Είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά εδώ σήμερα βρίσκεται μαζί μας ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουμε να τον συναντήσουμε υπό την ιδιότητα αυτή. Συνήθως έχουμε μια σύντομη παρουσίαση από αυτόν και μετά ακολουθούν ερωτήσεις, όπως κάνουμε συνήθως κάθε φορά που τον συναντάμε και τον γνωρίζετε πολύ καλά. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Τρισέ, προηγουμένως σας καλωσορίζω υπό την ιδιότητα του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο που εμφανίζομαι σε αυτή την επιτροπή σήμερα υπό την ιδιότητά μου σαν πρόεδρο ε, του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου του Αρμοδίου για το Συστημικό Κίνδυνο, για να εξηγήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω άλλωστε προβλέπεται στο άρθρο 5,4 του κανονισμού του, του Συμβουλίου μα αυτού, ε, πώ προτίθεμαι να εκτελέσω τα καθήκοντά μου. Τώρα είναι κρίσιμο είναι, πρέπει να το συγχαρούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη νέα εποπτική αρχιτεκτονική του και ότι χρησιμοποιεί μια ταχεία νομοθετική διαδικασία. Η μεταρρύθμιση δείχνει ότι η Ευρώπη μπορεί τελικά να αποδώσει. Στις σημερινές μου δηλώσεις επιθυμώ, στα γερμανικά συνεχίζει τώρα μετά από τα πολωνικά, τι σκοπεύουμε, ή μάλλον πώς σκοπεύουμε να θέσουμε τις βάσεις για την περαιτέρω εργασία του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Ο στόχος μας είναι να επιτύχουμε, ε, να επιτύχουμε εργασία και συνεργασία του Συμβουλίου ήδη από τον Μάρτιο που θα αφιερώσει την πρώτη αυτή συνεδρίαση σε ουσιώδη θέματα. Πρόκειται δηλαδή για τη δουλειά που ήδη έχει γίνει και για τις διάφορες αποφάσεις ε, που λάβαμε για να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή εντός των απαιτουμένων χρονικών περιθωρίων, την εύρυθμη λειτουργία της νέας αρχής ε, που, δημιούργησε η, που είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Συστημικού Κινδύνου. Ε, σε μια δεύτερη φάση θα αναφερθώ στην μακροπολιτική εποπτείας συνετής διαχείρισης του φορέα αυτού, καθώς και τις συστάσεις και τους συναγερμούς που θα γύρει στα πλαίσια το απαραίτητα των πολιτικών που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν θα τονίσω ότι αυτός ο φορέας ξεκινά τώρα τις δραστηριότητές του μετά την σύστασή του εδώ και 7 εβδομάδες στην εναρτήρια συνεδρίαση που έλαβε χώρα εδώ και 2 εβδομάδες. Επιπλέον, η εποπτεία, η μακροοικονομική συνετή διαχείριση είναι ένα τομέα πολιτική πράγματι οι συνάδελφοί μου και εγώ έχουμε πιστεί ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στη σύσταση του φορέα αυτού της Ευρωπαϊκή Επιτροπής Συντημικού Κινδύνου. Λοιπόν, στις 16 Δεκεμβρίου 2010 ε, ο νόμος που δημιουργεί αυτό το Συμβούλιο Συνδικού Κινδύνου, το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, ετέθησε ισχύ και ξεκίνησε η θητεία μου ω ε, ε, ως Προέδρου αυτού του φορέα. Ταυτόχρονα την ίδια μέρα, ο κύριος Μέρβιν Κίνγκ, ο οποίος είναι διοικητής τράπεζας της Αγγλίας, εξελέγει πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συνδικού Κινδύνου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στις 20 Ιανουαρίου του 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, είχε την ανακτήρια συνεδρίασή της και αυτή η συνεδρία αρχικά ασχολήθηκε με τη δημιουργία των θεμελίων τη βάσεω για το νέο φόρε αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ εκτενέστερε αποφάσει που λάβαμε εκείνη την ημέρα. Η Διευθύνουσα Επιτροπή αποτελείται από 14 μέλη, συμπεριλαμβανομένων 4 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που, του, Γενικού Συμβουλίου, που είναι και μέλη του Γενικού Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τραπέζη. Στι 20 Ιανουαρίου του 2011, ο κ. Μάρεκ Μπέλκα, διοικητή τη Narodowy Bank Polski, ο κύριος Μάριο Ντράγκη, διοικητής της Banca d'Italia, ο κύριος Αθανάσιος Ορφανίδης της ε, Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και ο Άξελ Βέμπερ, πρόεδρος της Deutsche Bundesbank, εξελέγησαν μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής για τρία χρόνια. Την ίδια μέρα, ο κύριος Στέφαν Ίγκβες, διοικητής της Φέριξες Riksbank, εξελέγει πρόεδρος της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής για μια τριετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εντολή που θα δινόταν σε αυτή την Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή. Η Εν Λόγω Επιτροπή θα παρέχει συμβουλές και βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική, στο φορέα μας και θα αναθεωρούμε τακτικά τι δημοσιονομικέ συνθήκε σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένε και τη εντόπιση συστημικών κινδύνων. Πιστεύω ότι η Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή μπορεί να διαρματίσει επίση σημαντικό ρόλο όσον αφορά την αναθεώρηση και ανάπτυξη μακροοικονομικών μέσων πολιτική για συνετή διαχείριση. Αντικυκλική ειδικά κεφαλουχικά ε, κεφάλαια για τη μετώπιση των κινδύνων ε, θα είναι ένα τέτοιο μέσο. Και τελείωσαν πρόσφατα δημόσιε διαβουλεύσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το θέμα. Τώρα, στρεφόμενο προ την Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύσει ε, μία, ένα διαγωνισμό για εξωτερικούς συμβούλους που θα πρέπει να διοριστούν σαν μέλη αυτής της επιστημονικής επιτροπής, συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής. Να πω μερικά λόγια όσον αφορά αυτό το συμβουλευτικό φορέα ε, για τον οποίο ενδιαφέρεται και έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον το Κοινοβούλιο. Λοιπόν, η προκήρυξη του διαγωνισμού ε, βρίσκεται στην ιστοσελίδα του φορέα μας και θα δημοσιευθεί αύριο σε όλες τις επίσημες γλώσσες ε, της επίσημες εφημερίδας. Ε, η δημοσίευση ε, αποτελεί την αφετηρία μιας ε, φάσεως επιλογής. Μετά από αυτό, οι υποψήφοι θα έχουν τρει εβδομάδε να υποβάλουν αίτηση. Στόχο είναι να προσελκύσουμε επιφανεί εμπειρογνώμονε και νομίζω ότι εδώ εκφράζουμε και τη βούληση του Κοινοβουλίου. Η εντολή αυτή τη Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή συμπεριλαμβάνει συμβολέ μάλλον όσον αφορά τον καθορισμό μεθοδολογιών για τον τοπισμό των κινδύνων και αξιολόγηση ενδεχομένων συνεπειών όσον αφορά την πραγματοποίηση αυτών των κινδύνων, όσον αφορά το σχεδιασμό και στάθμιση αποτελεσματικών εργαλείων για τη μακροοικονομική πολιτική συνετή διαχείριση, συμπεριλαμβανομένη και τη βελτιώσεω των υφισταμένων εργαλείων ή μοντέλων, καθώ και ανοιχτή, ανεξάρτητη και αναλυτική αναθεώρηση των μακροοικονομικών στρατηγικών συνετής διαχείρισης και των διάφορων λειτουργικών πλαισίων. Στη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης κατάρτισε τον εσωτερικό κανονισμό του φορέα μας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για Συνδικό Κίνδυνο και συμφώνησε όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα του 2011. Το πρόγραμμα προβλέπει τέσσερι περαιτέρω συνεδριάσει του Διοικητικού Συμβουλίου αυτό το έτο, τον Μάρτιο, τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο. Εν τέλει, η γραμματεία της Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου δημιουργήθηκε και έχει πάνω από 20 μέλη του προσωπικού από αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεω και με διαφορετικό επαγγελματικό ιστορικό και εμπειρία. Η ποικιλομορφία του προσωπικού συμβάλλει σε μια δημιουργική σύνθεση και σύνοψη ιδεών και την αποτελεσματική λειτουργία της γραμματείας, ούτως ώστε να βοηθηθεί ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Στημικού Κινδύνου να πετύχει τους στόχους του. Αυτή είναι μια σύντομη επισκόπηση τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε την έγκαιρη δημιουργία αυτού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Θα ήθελα τώρα να στραφώ για μια στιγμή προ το μέλλον, δηλαδή την μακροοικονομική ε, εποπτεία από πλευρά ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Ο κανονισμό δημιούργησε το φορέα αυτό σαν ανεξάρτητο όργανο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που είναι υπεύθυνο για τη μακροοικονομική ε, τη σκόπηση, έλεγχο μάλλον οικονομική διαχείριση του χρηματοπιστικού συστήματο εντό ενώσεω. Θα τονίσω τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο φορέα αυτό θα εστιαστεί όσον αφορά την πρόληψη και μείωση των συστημικών κινδύνων που απειλούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστικού συστήματο στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Υπότιτλοι Κάνοντα το αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε οριζόντιου κινδύνου σε όλα τα κράτη-μέλη, με ενδεχόμενο αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά την πραγματική οικονομία. Ο φορέα αυτό επίση μπορεί να ασχοληθεί με θέματα όσον αφορούν μια συγκεκριμένη χώρα, εάν αυτά τα προβλήματα δημιουργούν συστημική απειλή ή κίνδυνο για το χρηματοστατικό συστήματο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ε, μέσω επιδράσεω στα αλλα κράτη-μέλη και θα λαμβάνει υπόψη τι παγκόσμιε εξελίξει με ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, ε, ο φορέα αυτό έχει αποστολή, όπω το τόνισε και το Κοινοβούλιο, ε, μια, έναν ευρύ έλεγχο όσον αφορά τα μακροοικονομικά, όσον αφορά τη συνετή διαχείριση, που καλύπτει όχι μόνο τι τράπεζες, αλλά και διάφορου ε, φορεί διάφορους φορείς αγορές, προϊόντα και υποδομέ που ίσω να δημιουργούν προβλήματα και ανησυχίε όσον αφορά τη χρηματοστατική σταθερότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και τρίτον, η δραστηριότητα το, της, αυτού του φορέα θα θα αφορά ισχυρή συνεργασία μεταξύ 100 μελών και βασικό κομμάτι του φορέα θα είναι να συνδυάζεται η ανάλυση που παράγεται από του μικροεπόπτες και τι κεντρικέ ε, τράπεζε. Θα ήθελα να σα αναφέρω ότι η εναρτήρια συνεδρίασή μας ε, έδειχνε πολλέ υποσχέσει όσον αφορά αυτά τα θέματα. Τώρα ξεκινάμε τι μακροοικονομικέ ε, δραστηριότητε υποπτία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τιμικού Κινδύνου σε επιχειρησιακό επίπεδο. Συμφωνήσαμε στο επίπεδο του Διοικητικού Συμβουλίου να εξετάσουμε το στιμικό κίνδυνο στο χρηματοστικό σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ε, κάθε τρίμηνο. Ε, το Διοικητικό Συμβούλιο όμω μπορεί ίσω να μελετήσει και μακροπρόθεσμα διεθνωτικά θέματα που αφορούν την ε, δημοσιονομική χρηματοστική σταθερότητα, διότι ίσω να δημιουργήσουν κάποιου κινδύνου στο μέλλον. Οι συζητήσει του Διοικητικού Συμβουλίου προετοιμάζονται όπως αποφασίσετε εσείς από τη Διευθύνουσα Επιτροπή ε, του φορέα αυτού επί της βάσεως συνεισφορών όλων των ε, θεσμών που συμμετέχουν. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ε, αναφέρεται σε βασικού συστημικού κινδύνου που διαβλέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί τη βάση ε, τη αναλύσεω που προβάλλει όσον αφορά την ευρεία χρηματοστατική σταθερότητα. Η Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου θα χρησιμοποιεί και του δείκτες αυτού, του ποσοτικούς και ποιοτικού, καθώ και τα διάφορα αναλυτικά εργαλεία που υπάρχουν. Εκεί συμπεριλαμβάνουν ιδιαίτερα διάφοροι δείκτες για τη χρηματοστατική σταθερότητα, συστήματα έγκαιρη προειδοποίηση και δείκτε και μοντέλα ε, δυνατότητα επιμόλυνσης και διάφορες δοκιμές αντοχής για να αναδειχθούν περαιτέρω αναλυτικά μέσα για την υποπτία την μακροοικονομική συνετής διαχείρισης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και, τα, και κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο που αποκαλείται εμά από το Macro Regulation Supervision το οποίο ασχολείται με την ε, έρευνα στον αφορά τον τομέα της μακροοικονομικής διαχείρισης και η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου έχει μια εντολή να συμβάλλει σε ανατηλικές μεθοδολογίες ούτως ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται διάφοροι συστημικοί κίνδυνοι. Για να εξασφαλίζεται μια πολύ καλή ανάλυση των συστημικών κινδύνων, ε, σχεδιάζουμε να συλλέξουμε, να έχουμε μια διαδικασία συλλογή διαφόρων στοιχείων για ε, έλεγχο μακροοικονομικό συνετή διαχείριση που θα βασίζεται στα διάφορα δήματα που συμμετέχουν. Επίση, συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει δεδομένα για μακροοικονομικέ εξελίξει και όλα τα διαθέσιμα ε, στοιχεία για, του χρηματοστατικού συστήματο για μακροοικονομικού λόγου συνετή διαχείριση και οι ευρωπαϊκέ εποπτικέ αρχέ διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη συλλογή εποπτικών στοιχείων όσον αφορά τα ιδρύματα για τον Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Στιμικού Κινδύνου που κατά κανόνα θα, εξαφανί... θα εξετάζονται σε μαδοποιημένη μορφή. Όλε αυτέ οι πληροφορίε συμπληρώνονται από στοιχεία τη αγορά, από εμπορικά στοιχεία που παρέχονται από διάφορου συμμετέχοντε, καθώ και από διάφορε πληροφορίε που συλλέγονται για την αγορά από διάφορους, ε, διάφορα σημεία επαφή και διάφορου εμπλεκόμενου του ιδιωτικού τομέα. Και θέλουμε να εκδίδουμε συστάσει και προειδοποίησει όσον αφορά για δράσει που χρειάζονται για διόθεση καταστάσεω. Η Συμβουλευτική Τεχνική μας Επιτροπή θα ξεκινήσει να ερευνά ενδεχόμενα μέσα για την διαμόρφωση πολιτικής βάσει των οποίων ο φορέας μας μπορεί να κάνει συστάσεις. Όσον αφορά την προετοιμασία για προειδοποίησεις και συστάσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου θέλει να εντάξει όλη την αναγκαία τεχνογνωσία με τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο. Για αυτό το σκοπό, η Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή θα συμμετέχει σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο των προετοιμασιών και διάφορα και από τα διάφορα θεσμικά όργανα, διάφοροι εμπειρογνώμονε μπορούν να διδραματίσουν σημαντικό ρόλο σαν αφορά. Όπω αποφασίστηκε λοιπόν από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου ε, δεν έχει δεσμευτικέ εξουσίε. Ε, θα πρέπει να μιλά με πειθό και να δημιουργήσει αξιοπιστία με την πάροδο του χρόνου. Για τι συστάσει του φορέα μα θα πρέπει να υπάρξει μηχανισμό για να δίνει συνέχεια στι συστάσει επί τη βάση τη αρχή του συμμορφώσου ή εξήγησε. Είναι κάτι που προβλέπεται αυτό ο μηχανισμό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα αποφασιστικό ρόλο να διαδραματίσει σχετικά με αυτό το θέμα. Πιο συγκεκριμένα, εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου ε, δημοσιεύει τι συστάσει, το Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει τον πρόεδρο του φορέα αυτό να παρουσιάσει τι συστάσει και επίση που οποίου απευθύνονται προειδοποίηση θα μπορούν να συμμετάσχουν ανταλλαγή απόψεων. Όμω, αν οι συστάσει τελικά παραμείνουν εμπιστευτικού χαρακτήρα, ίσω θα πρέπει να συζητηθούν εμπιστευτικά σε προφορικέ συζητήσει που θα ε, διοργανώσει ο πρόεδρο του φορέα μα τουλάχιστον δύο φορέ ε, το χρόνο και κλεισμό των θερών. Αυτό είναι απόφαση δική σα. Με τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο τη Επιτροπή σα. Πιο γενικά, είμαι απόλυτα βέβαιο ότι το Κοινοβούλιο θα ακολουθήσει εκ του σύνεγγυ ε, το έργο τη Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή του Κίνδυνο και πολύ χαίρομαι που αποφασίσατε να θα ετησίως για να παρουσιάζουμε την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ίσως να ζητηθεί να ερχόμαστε σε ακροάσεις ενώπιον των αρμοδίων επιτροπών. Ε, εγώ περιμένω μια πολύ ε, θετική διάδραση ε, τους επόμενους μήνες. Θα ήθελα να κλείσω διαβεβαιώνοντάς σας ότι ο κύριος Μέρβιν Κίν, ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο δεύτερος αντιπρόεδρος ε, που είναι από, την Ευρωπαϊκ... από τις Ευρωπαϊκές Αποπτικές Αρχές και εγώ μαζί με όλους τους συναδέλφους που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε στη σημαντική αποστολή που η Ευρώπη μας ανέθεσε, που ανέθεσε στο νέο μας αυτό θεσμό. Θα εργαστούμε για να εντοπίσουμε τους σωστούς κινδύνους και να προβούμε στη δέουσα ανάλυση και να δώσουμε τις αναγκαίες συστάσεις και προειδοποίησεις που μας ζητήσατε να επεξεργαστούμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα προχωρήσουμε σε ερωτήσεις και απαντήσεις. Παρακαλώ σε χρονικά όρια πέντε λεπτών και εγώ είμαι υποχρεωμένη να τηρώ τον χρόνο. Ζαν Πολ Γκοζές, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα χαίρομαι, εκφράζω την ικανοποίησή μου για την σοφία των όσων ε, έχουν συντάξει οι ε, συνάδελφοί μου συντάξτες της γνωμοδότησης. ώστε ο πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας να είναι και πρόεδρο του Συμβουλίου Συστημικών Κινδύνων, αποφεύγοντα έναν θεσμικό κίνδυνο, ένα θεσμικό διάλογο μάλλον για τον κίνδυνο τη αποδυνάμωση τη Ευρωπαϊκή Εποπτεία. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Κατά τα λοιπά γνωρίζετε ότι τι ημέρε, τις προηγούμενες ημέρε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φροντίσαμε ώστε να μην αποδυναμωθούν τα όσα επιθυμούσαμε να διαθέτει ως εξουσίες η ε, αρχή μέσα στα πλαίσια βέβαια του νομοθετικού πλαισίου που την ε, ε, ρυθμίζει. Η δήλωση του Επιτρόπου αλλά και της Ουγγρικής Προεδρίας τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας μας επέτρεψαν να διαθέτουμε ορισμένε σχετικές διασφαλίσεις. Θα σας ρωτήσω πώς βλέπετε στο μέλλον τη σχέση σας με τις τρεις αρχές εποπτείας των οποίων οι πρόεδροι μόλις ορίστηκαν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Yes, yeah, yeah, yeah. You can start. Merci, beaucoup de, de Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Συγχαίρω πρώτα τους επικεφαλείς των αρχών εποπτείας που όπως είπατε μόλις διορίστηκαν όταν διεξαγάγαμε την πρώτη μας συνεδρίαση εγγενείων δεν τους γνωρίζαμε ακόμα, δεν τους είχαμε ακόμα. Θεωρώ πάντως ότι η συνεργασία που θα έχουμε όπως την επιθύμησε άλλωστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συνεργασία αυτή θα είναι και στενή και εμπιστοσύνη. Έχουμε ήδη με τη στενή συνεργασία των αρχών διεξαγάγει την πρώτη αυτή συνεδρίαση και εντυπωσιάστηκα πραγματικά από το γεγονός ότι τόσο σημαντικά έγγραφα, όπως για παράδειγμα ο κανονισμός των εργασιών μας, που ασφαλώς περιέχουν πολλές λεπτομέρειε και είναι ιδιαίτερα περίπλοκα έγγραφα, είναι εκφίσω έτσι. Πάντως συντάχθηκαν μέσα σε πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας. Είμαι πεπισμένος ότι η συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου συστημικού κινδύνου και των αρχών εποπτείας και σε ό,τι αφορά την συλλογή δεδομένων και πληροφοριών και την αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων τις όσες διατομιακές ε, ενέργειες θα πρέπει να αναλάβουμε θεωρώ ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Οι πρώτες επαφές που διεξαγάγαμε έδειξαν πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να διασταυρώνουμε τις αναλύσεις μας από όλες τις πλευρές, ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή επισκόπηση, η ευρύτερη δυνατή εικόνα του συστημικού κινδύνου. Νομίζω ότι μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα είναι ε, αγαστή η συνεργασία. Ακόμα βέβαια δεν έχει αρχίσει, θα σας τα πω όταν θα επανέλθω την επόμενη φορά να σας δω. Σας ευχαριστώ. εξ ονόματος τώρα του, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η νομισματική μάζα αυξάνει ε, σε όγκο. Αυτό θέτει δύο προβλήματα. Αφενός στην αγορά ενεργητικών υπάρχει ένας πληθωρισμός που θέτει ένα συστημικό κίνδυνο νέων ε, ότι μπορεί να, ξα, ξανασκάσει κάποια φούσκα. Πώς το βλέπετε εσείς μέσα στα πλαίσια των νέων σας καθηκόντων. Και δεύτερο, εάν φαίνεται αυτό να έχει μια νομισματική διάσταση στην πραγματική οικονομία, προφανώς δεν είναι έτσι συνδέεται πολύ περισσότερο με την έκρηξη των τιμών των πρώτων υλών καθώς και του ε, μισθολογικού κόστους. Μείωση των επιτοκίων προφανώς δεν θα είχε κανένα νόημα εφόσον δεν είναι νομισματικού χαρακτήρα ο πληθωρισμός. επόμενες, τους επόμενους μήνες, εάν επιβεβαιωθεί η αύξηση αυτή του πληθωρισμού, θα αυξήσετε τα επιτόκια. Γνωρίζοντας βέβαια ότι η ανάκαμψη είναι ακόμα πολύ εύθραυστη. Ε, ε, Κοιτάξτε, κύριε και κύριοι, η ερώτηση είναι ερώτηση για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και ναι, ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ευχαρίστως αν ε, με καλείτε ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να σας απαντήσω και να σας εξηγήσω, αλλά ως πρόεδρος του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου έχω την αίσθηση ότι πρέπει να διακρίνουμε τα πράγματα. Τα δύο όργανα δεν πρέπει να μπερδεύονται καθόλου. Υπάρχει η συνθήκη του Μάστριχτ από τη μια μεριά, υπάρχει από την άλλη μεριά η νομοθεσία που δημιουργήσατε εσεί. οπότε θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και να μην μπερδεύουμε τις δύο αυτές αρμοδιότητες και τις δύο ακροάσεις. Συμφωνείτε κύριε Πρόεδρε, θέλω να με καθοδηγήσετε σε αυτό. Συγγνώμη, λέει ο Ευρωβουλευτής, το πρώτο δεν είναι τέτοιο θέμα. Η Πρόεδρος. Είναι πολύ σημαντικό όντω να μην μπερδεύουμε εδώ πέρα τα δύο είδη διαλόγων που έχουμε με τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τη μια και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου από την άλλη. Είναι πολύ σημαντικό Πολλέ φορέ. Μα το υποσχέθηκαν ότι θα υπάρχει διάκριση ανάμεσα στα δύο. Και εγώ το φαντάστηκα ότι τη δυσκολία θα την είχαμε και μάλιστα είχα σκεφτεί ότι εγώ θα έχω πιο πολύ αυτή τη δυσκολία παρά ευρωβουλευτέ. Εν πάση περιπτώσει, μήπω υπάρχει κάποιο τμήμα τη ερώτηση του Ευρωβουλευτού που κύριε Τρισέ θα μπορούσατε να απαντήσετε υπό την ιδιότητά σα ω πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Ο κύριο Τρισέ. Μπορώ να επαναλάβω αυτό που είπατε για την νομισματική μάζα. Είναι θέμα αριθμών. Η νομισματική μάζα, το M3, είναι κάτι που παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε όμως με ιδιαίτερη προσοχή και τα συνθετικά του. Αλλά αυτή η νομισματική μάζα αυξάνεται λιγότερο γρήγορα από ότι το καθάριστο ΕΠ. Οπότε νομίζω ότι παρακολουθείτε και άλλους δείκτες εκτός από το M3. Αυτό. Δεν έχω, θέλω να πω τίποτα παραπάνω επ' αυτού. Ευχαριστώ. Το επόμενο ερώτημα όσον αφορά την Άλτε. Η Σιλβί Γκουλάρ που ήταν η συγγήτρια για το Συμβούλιο του Συστημικού Κινδύνου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχεί διότι έγινε συλλογική δουλειά εδώ με όλους τους σκιώδεις που μου περιτριγύρισαν, ούτω ώστε σήμερα να είστε μπροστά μα υπό αυτή την ιδιότητα. Ένα σχόλιο και ένα ερώτημα. Το σχόλιο αν αναφερθείτε αναφερθήκατε εμά στην Επιστημονική Επιτροπή. Ξέρετε ότι και αυτό είναι μια καινοτομία που προέρχεται από το Κοινοβούλιο και δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό το φορέα και σε ευχαριστώ που το υπογραμμίσατε, διότι πρέπει να υποθεί αυτό, ότι η φιλοδοξία μας στον τομέα αυτό ήταν να επιτρέψουμε να περιτριγύριζεστε από συμβούλους ε, παγκοσμίου επίπεδου. Ε, θέλουμε το μεγαλύτερο δυνατό άνοιγμα και επίσης να υπάρχουν όλοι οι τομείς, να εκπροσωπούνται οι περισσότεροι δυνατοί Λοιπόν, ρίξατε τα δίκτυα σα δεν ξέρω τι ψάρια θα πιάσετε. Ε, όμως ε, παρακολουθούμε. Το ερώτημα είναι αυτό που θα συμβεί στον τομέα του τραπεζικό και τον τρόπο με τον οποίο υπό την έποψη συστημικού κινδύνου θέλετε να συνεργαστείτε ε, με τις διάφορες αρχές της τραπεζικής για τις επόμενες δοκιμές αντοχής και τους ελέγχους που θα πρέπει να γίνουν στον αφορά τον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό τομέα. Ευχαριστώ και τον προτέρων κύριε Πρόεδρε. Okay. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως είπα και πριν από λίγο, ακολουθούμε το γράμμα των όσων εσείς αποφασίσατε όσον αφορά την Επιστημονική Επιτροπή, αλλά και το πνεύμα των όσων αποφασίσατε. Βλέπετε η διαδικασία τώρα ξεκινάει, προχωράει, δεν χάνουμε όμως χρόνο. Προσπαθούμε να συμφωνήσουμε και ξεκινήσαμε ήδη από την πρώτη μας συνεδρίαση. Οπότε εφόσον θέλετε, ευχαρίστως θα αναφέρω τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής εκδήλωσης ενδιαφέροντος που προκηρύξαμε. Όσον αφορά τις σχέσεις μας τώρα με τις τραπεζικές αρχές, όλος ιδιαίτερος. Οι πρώτες επαφές που είχαμε στην αρχική συνεδρίαση της Επιτροπής μας ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αυτό που θα είναι η τραπεζική αρχή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανέφεραν τον τρόπο με τον οποίο ξεκινούν την άσκηση των δοκιμών αντοχής. Όπως είπα και πριν από λίγο, η Τεχνική Συμβουλευτική μας Επιτροπή θα ασχοληθεί με αυτή την πτυχή που είναι όντω σημαντική. Νομίζω ότι μπορώ να σας πω πως η συνεργασία ανάμεσα στα διάφορα όργανα που είναι αναγκαία γίνεται προς το παρόν μέσα σε ένα πολύ εργαστό πνεύμα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Είναι όμως μια σημαντική δουλειά όπως καταλαβαίνετε που προχωράει και που σίγουρα χρειάζεται να επιδείξει ο καθένας μας ιδιαίτερο επαγγελματισμό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους του ECR τώρα παρακαλώ. Ο κύριος Έπινγκ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ορισμένοι ηγέτες Ευρωπαίοι ε, πρότειναν ε, περικοπές, ε, πρότειναν οι επενδυτές περισσότερο τις απόλυ... να αναλάβουν περισσότερο τις απώλειες ήδη επενδυτές παρά άλλοι που έχουν χάσει. Αυτό όμως μήπως θα οδηγήσει σε έκθεση των ε, άλλων θεσμικών φορέων. Αυτό δεν θα οδηγήσει σε ένα συστημικό κίνδυνο. Εξαρτάται βέβαια, όταν είπαν περικοπέ, ε, χρησιμοποιεί ο μιλητή την έκφραση να κόψουν τα μαλλιά, τις τρίχες. Μήπως όμως τελικά εξαρτάται από το πόσα μαλλιά διαθέτει κανείς και αν έχει λίγα τελικά δεν θα του μείνει τίποτα. Έτσι το λένε. Κούρεμα. Και εφόσον είσαστε και πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν και ξέρω ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο εδώ, πείτε μου έστω ω πρόεδρο του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, εσεί πώ βλέπετε αυτό το κούρεμα που προτείνανε. Έχετε μια άποψη, δύο απόψει, μια που έχετε και δύο διαφορετικέ ιδιότητε. Για πείτε μα. Με τα δικά σας τα κριτήρια εγώ δεν θα έπρεπε να ανησυχώ και πολύ, μια που έχω μαλλί αλλά επιτρέψτε μου όμως να σας εξηγήσω περισσότερο. Πρώτα απ' όλα, έχουμε προγράμματα για την Ελλάδα, τα οποία έχουν εγκριθεί από τη διεθνή κοινότητα, από το Διεθνές Μεσονατικό Ταμείο, από όλο τον κόσμο και έχουν εγκριθεί και από την ε, Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις κυβερνήσεις στο βαθμό που συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα αναπροσαρμογής. Το μήνυμα είναι απλό. Πρέπει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα, όπως γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις μέχρι τώρα. Εφαρμογή του προγράμματος. Αυτό είναι το μήνυμα που έχουμε και εμείς για την ελληνική κυβέρνηση. Στην Ιρλανδία ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Και εκεί Εγκρίθηκε ένα πρόγραμμα από τη διεθνή κοινότητα, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Μαθητικού Ταμείου, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρηματοδοτείται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφαρμόστε το πρόγραμμα, εφαρμογή του προγράμματος. Το πρόγραμμα δεν προκαταλαμβάνει αυτά που λέτε εσείς, εφαρμογή του προγράμματος χρειάζεται. Για να υπάρξει ανάκτηση της αξιοπιστίας πρέπει κανείς να αποδείξει ότι εφαρμόζει το πρόγραμμα να είναι πιστικό αυτό ότι κάθε τρίμηνο τηρεί το πρόγραμμα, το εφαρμόζει σωστά. Και κοιτάμε σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το πρόγραμμα αυτό. Τώρα επιτρέψτε μου να προσθέσω μια τελευταία παρατήρηση μόνο. Οι σύγχρονες αγορές είναι φτιαγμένες με επενδυτές οι οποίοι έχουν αντοχές μεγάλες ή λιγότερο μεγάλες. Η πρώτη, η ιδιωτικό τομέα, για παράδειγμα, χάνει χρήματα όταν ε, θέσουμε σε εφαρμογή το χοντροκούρεμα, αυτό στο οποίο αναφερθήκατε. Οι άλλοι κερδίζουν χρήματα. Οπότε αυτό πρέπει κανείς να έχει υπόψη του όταν ε, σκέφτεται αυτό το ζήτημα. Το μήνυμα πάντως είναι εφαρμόζουμε το σχέδιο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Πασκάλ Καμφά από τους Πρασίνους, παρακαλώ, από την ομάδα των Πρασίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρου των Πρασίνων, ε, χαιρόμαστε που δημιουργήθηκε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Πρώτα απ' όλα, διότι θα είναι το μόνο όργανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχει την ευθύνη να ελέγχει τα ιδιωτικά χρέη. Βλέπουμε όμω τη συζήτηση που γίνεται για το σύμφωνο σταθερότητα και από την ιστορία τη πρόσφατη κρίση, βλέπουμε ότι όταν επικεντρωνόμαστε υπερβολικά στο δημόσιο χρέο είναι μάταιο γιατί ένα μεγάλο μέρο του σημερινού δημοσίου χρέου προέρχεται από το ιδιωτικό χρέο. γιατί αντικαθιστά το ιδιωτικό χρέο. Αυτό το βλέπουμε και στην Ιρλανδία και στην Ισπανία και όχι μόνο. Συνεπώ. η ευθύνη που αναλάβατε είναι σημαντική και θέλουμε εμεί να ξέρουμε εσεί. Πώ θα αντιθέσετε σε εφαρμογή. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις έχω. Η πρώτη που έχει να κάνει και με εκείνη του συναδέλφου από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Και σας ρωτάω υπό την ιδιότητά σας Προέδρου του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Ένας από τους τρόπους για να μειωθεί, ή να μειωθεί ο κίνδυνος για φούσκες, το ιδιωτικό χρέο δηλαδή, είναι η αύξηση των επιτοκίων. Συνεπώ, ο Ζαν Κλοντ Κρισέ, πρόεδρο του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, θα προτείνει τέτοιε συστάσει στο Ζαν Κλοντ Τρισέ υπό την ιδιότητα του πρόεδρου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση των επιτοκίων. Αν μα πείτε πω όχι, γιατί θεωρείτε ότι δεν είναι αυτό που πρέπει να γίνει για να μειωθεί ο συστημικό κίνδυνο, τι θα κάνετε, τι εργαλείο θα χρησιμοποιήσατε. Πολλέ φορέ είπατε στην εισαγωγή σα ότι πρόκειται για εργαλεία. Ε, μακροπροληπτικής εποπτείας. Αλλά δεν μα αναφέρατε ποια είναι αυτά. Οπότε αν είναι δύσκολο για εσά να αναλάβετε κάποια δέσμευση για το μέλλον, μπορείτε να μα πείτε κατά το παρελθόν τι θα κάνετε εσεί αν ήσασταν πρόεδρο του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου νωρίτερα για να αποφύγετε τι φούσκε ιδιωτικού χρέου στην Ιρλανδία και την Ισπανία. Τρισέ. Ευχαριστώ πολύ για να διευκρινίσουμε τα πράγματα όσο γίνεται πιο ξεκάθαρα. Η συνθήκη του Μάστριχτ ζητάει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προσφέρει σταθερότητα τιμών. Αυτή είναι η πρώτη εντολή που έχει. και να στηρίξει στη συνέχεια τις διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές. Η πρώτη όμως εντολή που έχουμε είναι σταθερότητα τιμών. Το δόγμα μας είναι πολύ απλό τα στάνταρ μέτρα μας, δηλαδή επιτόκια που βρίσκονται και στον πυρήνα των ε, στάνταρ μέτρων, καθορίζονται έτσι ώστε να υπάρχει σταθερότητα τιμών μεσοπρόθεσμα. Οπότε από αυτή την άποψη, υπό την ιδιότητα του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με ικανοποίηση μπορώ να πω μέχρι τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς διαπιστώσαμε ότι τα ε, πρώτα χρόνια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά το σύνολο της Ευρωζώνης έχουμε σταθερότητα τιμών κάτω από 2% ετησίως 1,97% για την ακρίβεια, κάτω από 2% λοιπόν. Και αυτό ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τον ορισμό που δίνουμε εμείς στη σταθερότητα τιμών. Μπορώ επίσης να πω και θα με ελέγξετε κι εσείς γι' αυτό, ότι όταν αποφασίστηκε η συνθήκη του Μάστριχτ και επικυρώθηκε από όλες τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Η βαθιά πεποίθηση των Ευρωπαίων ήταν σταθερότητα τιμών σημαίνει αναγκαία προϋπόθεση για την εφόρο για την απασχόληση και για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αναγκαία λοιπόν προϋπόθεση αλλά όχι και επαρκής από μόνη της. Διότι χρειάζεται να συνοδεύεται και από ε, δημοσιονομικές πολιτικές που να είναι σόφρονες, χρειάζονται και διευθυντικές πολιτικές και χρειάζονται και ένα σωρό άλλες ε, μακροοικονομικές πολιτικές, ενδεχομένως μακροπροληπτικές, ώστε να φροντίσουμε να έχουμε και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την οικονομική σταθερότητα ε, και την ανάπτυξη. Άρα είναι αναγκαία συνθήκη, αλλά δεν φτάνει από μόνη τη. Να ποια είναι η σχέση τη νομισματική πολιτική λοιπόν και τη Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου. Έρχομαι τώρα στο απευθεία ερώτημα που μου θέσατε. Είμαστε στις αρχέ μας. Σημαίνει ότι ετοιμάζουμε τον κατάλογο με τα διάφορα εργαλεία, τα διάφορα μέσα μακροπροληπτικής εποπτείας που έχουμε για να αποφύγουμε συστημικούς κινδύνους. Πολλά από αυτά τα μέσα εξετάζονται αυτή τη στιγμή από τη Συμβουλευτική μας Επιτροπή. Υπάρχει το long to value ratio, για να αναφερθώ στη δικιά σας συγκεκριμένη περίπτωση που είπατε πώς μπορούμε να αποφύγουμε τη δημιουργία ε, φούσκας ξανά. Ε, υπάρχουν όλα αυτά που έχουν συζητηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο για τα αντικυκλικά μέτρα που αποφεύγουν τις κρίσεις και που μας επιτρέπουν με διάφορα μέτρα να πλαισιώνουμε τους κινδύνους ακριβώς όταν θα κινδύνευαν να δημιουργήσουν φούσκες και συστημική κατάρρευση. Όλα αυτά τα καταγράφουμε τα περιλαμβάνουμε σε ένα κατάλογο σιγά σιγά. Έχουμε μεγάλη δυνατότητα ανάλυσης, μία εντελώς πολύπλευρη οπτική μια που προερχόμαστε από διάφορους τομείς και έτσι θα καταλήξουμε σε συστάσεις και σε προειδοποίησεις. Όμως δεν είμαστε εμείς που θα αποφασίσουμε. Γιατί δεν είναι αυτό που θέλετε εσείς. Αλλά νομίζω ότι το Συμβούλιο θα μπορεί να επηρεάσει πολύ εφόσον έχει τις σωστές συστάσεις, έχει καταλήξει σε σωστές συστάσεις. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Θυμάμαι όταν δημιουργούσαμε αυτό το Συμβουλίο Κινδύνο ότι είχαμε κάποια συζήτηση για τα συγκρούμενα συμφέροντα. Δηλαδή, πρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τη της Επιτροπής αυτής του Δημικού Κινδύνου. Ε, θα ήθελα να σας υποψηφίσω από το ερώτημα, να δω αν έχετε άποψη από αυτού, θα το κάνω. Γι' αυτό έχουμε ξεχωριστέ ακροασει. Λοιπόν, μην προσπαθήσετε να είστε έξυπνο και να δημιουργείτε δύσκολε καταστάσει. Εδώ δεν είναι κάτι στη διαδικασία ε, δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο γιατί δεν μπορούμε καν τελειώσουμε τον κατάλογο τον κανονικό που έχουμε ετοιμάσει για την υποβολή ερωτήσεων διότι έχουμε τρεις ή τέσσερις θέσεις για ερωτήσεις ακόμα στη θέση μας. Το επόμενο ερώτημα εκ μέρου του ΕΛΚ ο Μπέρκαρτ Μπάλτς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μια σύντομη ερώτηση. Μιλήσατε προηγουμένως για haircuts, για κουρέματα. Τώρα προτείνεται επαναγορά των ομολόγων από τις ενδιαφερόμενες χώρες. με δανεισμό σε Ελλάδα και Ιρλανδία των χρημάτων για να μπορέσουν να ξανααγοράσουν τα ομόλογα αυτά. Εγώ δεν θα σχολιάσω, αλλά αυτό το σενάριο μας οδηγεί σε ένα άλλο ερώτημα το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ως EASB και FAF πώς θα συνεργαστείτε στο μέλλον. Διεξάγεται ήδη η συνεργασία και ως πρόεδρος του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου εσείς ποιο ρόλο θα παίξετε στη συνεργασία αυτή. Thank you very much indeed. Απάντηση του πρόεδρου Το ερώτημα είναι ανοιχτό. Σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Είναι σαφές ότι η σταθερότητα της ζώνης ευρώ στο σύνολό της συστημικά είναι πάρα πολύ σημαντική και για τους 27. Μην λησμονείτε ότι ε, το Συμβούλιο εργάζεται και για τους 27 και είπαμε θα εξετάσουμε ποια μπορεί να είναι τα συστημικά στοιχεία και για τις 27 ε, χώρες μέλη. Γιατί από μία χώρα μπορεί να ξεκινήσει μία μόλυνση και των υπολείπων. Αυτό ασφαλώς είναι ένα θέμα το οποίο θα το εξετάσουμε. Μέσα στα πλαίσια τώρα του Συμβουλίου του ESAB όσο πιο σταθερή είναι η κάθε μία από τις συνιστώσεις των 27 τόσο το καλύτερο για το σύνολο των 27. Βέβαια δεν θέλω να προκαταλάβω τίποτα. Θα καθίσουμε να σκεφτούμε σοβαρά και σε βάθος ακριβώς αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Ελίζα Φερέιρα από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα πρώτα σας εύχομαι καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας και μία ερώτηση πάλι σχετικά με τα κουρέματα τις περικοπές αυτές για λόγους ασφαλείας. Μιλούν εδώ για αναρρύθμιση του χρέους ορισμένων χωρών. Δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα την τραπεζική, τραπεζική κρίση στην Ευρώπη. Θεωρείτε ότι η αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων διεθνών τραπεζών που είναι τόσο μεγάλες ώστε να μην επιτρέπεται να πτωχεύσουν, να μην μπορούν να πτωχεύσουν, θεωρείτε ότι η αντιμετώπιση αυτή ήταν μέχρι τώρα ορθή. Θα προχωρήσουμε σε μια ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή εξυγίανση των τραπεζών. μιλούν και για κινδύνους εποπτικούς. Πώς το βλέπετε αυτό σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την, τον εντοπισμό ανισορροπιών μέσα, ανάμεσα στις διάφορες οικονομίες. Το άλλο για την αναπροσαρμογή των μισθών θα έχει κάποια επίπτωση στις οικονομίες. Είναι δηλαδή μια κάποια λύση για την αντιμετώπιση της χρέωσης των χωρών. Ευχαριστώ για την πρώτη σας ερώτηση για τα κουρέματα συνολικά. Είπα ήδη όσον αφορά τα δημόσια χρέη. Είπαμε ότι έχουμε σχέδια, τα σχέδια αυτά πρέπει να εφαρμοστούν, να εκτελεστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όπως συνέβη σε όλο τον κόσμο. Και Κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό να μην προκαλέσουμε σύγχυση. Τα σχέδια αυτά έχουν εγκριθεί και εφαρμόζονται. Και αναμένω ότι η υπόθεση εργασίας της διεθνούς κοινότητας πλέον, όχι μόνο της ευρωπαϊκής, που έχει δείξει την ικανότητά της να προσαρμόζεται, σταδιακά θα γίνει και πιστική. Για την δεύτερη ερώτηση σας τώρα, για το δεύτερο πακέτο διακυβέρνησης. Το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου δεν το έχει εξετάσει. Είναι ίσως μια απάντηση βασισμένη στην κοινή λογική. Να πούμε ότι εφόσον προκαλούνται βελτιώσεις στην διακυβέρνηση κάθε μιας από τις συνιστώσεις των 27, κάθε μιας από τις χώρες των 27, τότε θα είναι καλό αυτό για την συστημική σταθερότητα και των 27. Αυτό είναι λογικό, αλλά το βλέπετε και εσείς αυτό το πράγμα, τα εξετάζετε και εσείς, άλλωστε πρόκειται να λάβετε μια πολύ σημαντική απόφαση στον διάλογο που διεξάγεται με το Συμβούλιο, με τις κυβερνήσεις. Ελπίζω πολύ, αυτό θα πω μόνο, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και πιο ειδικά η Επιτροπή σας θα δείξει ατσάλινη θέληση να προχωρήσει προς τα εκεί, γιατί Ο μέγας κίνδυνος προκύπτει από την ανεπαρκή διακυβέρνηση. Αυτό είναι ένα δίδαγμα το οποίο οφείλουμε να αντλήσουμε από την πρόσφατη εμπειρία μας. Τα ξέρετε καλύτερα και από μένα τι ακριβώς γίνεται, γιατί εσείς βρισκόσαστε μέσα στην καρδιά της λήψης των αποφάσεων. Για το τελευταίο θέμα που δείξατε, απάντησα στο sovereign debt στην πρώτη μου απάντηση, στο δημόσιο χρέος δηλαδή. Τώρα για το ότι οι ορισμένες τράπεζες είναι πολύ μεγάλες για να πτωχεύσουν. Αυτό απευθύνεται ε, απευθείας ε, στις τράπεζες, όντως. Διεξάγουμε στο παγκόσμιο επίπεδο μια πολύ σημαντική ε, συζήτηση για το νέο διαρκές καθεστώς, όχι για τώρα. Έχουμε τι διάφορε προφυλάξει του παγκόσμιου επίπεδου, έχουμε την Βασιλεία 3. Τι κάνουμε με του θεσμού αυτού που τα σύφη αυτά που είναι συστημικά, ε, συστημικά επηρεάζουν. Δεν μπορεί εδώ να δώσει μια απάντηση, για παράδειγμα, μόνη της, να δώσει μια απάντηση μόνη στους Ηνωμένε Πολιτείε, ούτε εμείς μόνοι μας. Διότι εξορισμού ασχολούμαστε με οργανισμούς πραγματικά διεθνείς και καμιά φορά παγκόσμιους, παγκόσμιας δραστηριότητας. Γίνεται πρόοδος, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι δεν θα πρέπει να ξαναβρεθούμε πάλι μπροστά σε μια δραματική κατάσταση όπως εκείνη που βρεθήκαμε μετά την κατάρρευση της τράπεζας Lehman Brothers. Πρέπει επίσης να πούμε ξεκάθαρα ότι πρέπει να προλάβουμε και εφόσον κάτι αποδειχθεί αναπόφευκτο, να έχουν δηλαδή μείζωνα προβλήματα αυτοί οι μεγάλοι συστημικοί οργανισμοί, να, μπορεί, να, να έχουν προβλήματα μεν, αλλά χωρίς να συμπαρασύρουν ολόκληρο το παγκόσμιο σύστημα. Να υπάρχει ένας διαμεθοριακός μηχανισμός δηλαδή επίλυσης των προβλημάτων αυτών και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Βολφ Κλίνς. Εδώ είμαι κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, νέα καθήκοντα αναλαμβάνετε τώρα και θα χρειαστείτε λίγους μήνες ίσως μέχρι να μπορείτε να μας πείτε τα πρώτα πράγματα ξεκάθαρα. Τον Μάρτιο όμως, λίγη θητεία σας, θεωρείτε ότι θα μπορέσετε μέχρι τότε να δώσετε ξεκάθαρες διαπιστώσεις για συστημικούς κινδύνους. Για παράδειγμα, ορισμένες ε, τράπεζες στην χώρα μου, τη Γερμανία, όπου υποψιάζουμε ότι έχουν διάφορους σκελετούς στα ντουλάπια τους, για να το πω έτσι. Προ ε, καιρού είχαμε ακούσει τον συνάδελφό μας Γκάι Μίτσελ, ο οποίος μας έλεγε, προ καιρού λέω τώρα έτσι, προσοχή, γίνεται, πάει να γίνει φούσκα των ακινήτων στην Ιρλανδία. Ωστόσο δεν λάβατε θέση τότε. Τι μου δίνει εμένα την ασφάλεια ότι ως πρόεδρος του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου θα είσαστε σε θέση να διείδετε έγκαιρα, να προβλέψετε έγκαιρα τον κίνδυνο αυτό και να λάβετε μέτρα για να τον αποφύγετε. Προβλέπω ότι όταν δεξαχθεί η πρώτη συζήτηση εντός του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου με θέμα το συστημικό κίνδυνο να μπορέσω να ενημερώσω. Θα δούμε κατά πόσο θα συζητηθεί δημοσία ή θα θεωρήσουμε ότι θα πρέπει να έχουμε σε άμεση επαφή μαζί σας κυρία Πρόεδρε. Αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά θα ξεκινήσουμε προσπάθειες ήδη. Είχαμε την εναρκτήρια συνεδρίασή μας, αλλά στην επόμενη συνεδρίαση θα μπούμε στις πλήρες εργασίες μας. Όπως είδατε θα έχουμε τρεις συνεδριάσεις στις οποίες θα συμμετάσχω πριν αποχωρήσω από τη θέση μου του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κατά συνέπεια σαν Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Για το ερώτημά σας, που ε- σε πρώτερες ακροάσεις με ρωτήσατε ποια θα είναι νομισματική πολιτική. Ξέρετε ότι αν είχαμε προσαρμόσει την νομισματική μας πολιτική, μη λαμβάνοντα υπόψη τα εκατομμύρια ανθρώπους στο σύνολό τους, αλλά Γερμανία ή Ιρλανδία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν θα είχαμε πετύχει σταθερότητα τιμών, ε, θα ήταν η διαφορετική κατάσταση. Άρα πρέπει να προσαρμόσουμε την νομισματική μας πολιτική λαμβάνοντας υπόψη μια τεράστια ενιαία αγορά με ένα νόμισμα όπου έπρεπε να προσέξουμε ποια θα είναι η συνετή διαχείριση σε χώρες κυρίως που απολάμβαναν αυτή την φούσκα έπρεπε, ε, έπρεπε να δούμε τι γίνεται με αυτούς τους διάφορους ε, φορείς επενδύσεων και τι γίνεται με τη φορολογική πολιτική. Ακόμα και αν τότε φαινόταν ότι η προσέγγιση ευθυγραμμιζόταν με τις απαιτήσει του Μάστριχτ. Ένα από τα μαθήματα που πήραμε από την κρίση ποιο ήταν ότι πρέπει κανείς να αποχωρήσει πιο πέρα, να καταλάβει πολύ καλύτερα τι είναι διαθροτικής μορφής. Αν είσαι σε περίοδο ακμής, είναι πολύ εύκολο ε, να πληρεί κανείς τα κριτήρια του Μάστριχτ. Και προς τις δύο κατευθύνσεις λοιπόν. Άλλες πολιτικές. Πιο συγκεκριμένα φορολογική πολιτική. Και συνετή διαχείριση ε, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά. Και όσον αφορά το δεύτερο θέμα, είμαστε στον τομέα που είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας. Όχι μάλιστα, συγγνώμη, στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Η Πρόεδρος, έχουμε χρονικό πρόβλημα, διότι η Γραμματεία ήταν αισιόδοξη όσον αφορά το πόσε ερωτήσει θα μπορούσαμε να καλύψουμε. Θα ακούσω και τι τρει από τι επίσημε ερωτήσεις. Άστριτ, Άντολιν και Βένα Λάγκεν. Παρακαλώ να είναι σύντομε οι ερωτήσεις σας και ο κύριος Τρισέ θα προσπαθήσει να απαντήσει μετά σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ, λέει κυρία Λούλινγκ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Τρισέ, γνωρίζω κάπως ε, αυτή τη θέση σας που έχετε δύο ιδιότητες. Ε, ήθελα να ξέρω λοιπόν αν η κρίση του κρατικού χρέους που σας ανησυχεί καθημερινά εδώ και μήνες σαν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι και ένα θέμα που ανησυχεί ιδιαίτερα Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με το μικρόφωνο της κυρίας Λούλινγκ. Euh. Ε, πρόεδρε, ερώτηση, λέει η κυρία Λούλινγκ. Σαν πρόεδρος της Επιτροπής για το Συστημικό Κινδύνο, αν το κρατικό χρέος σας απασχολεί ιδιαίτερα, πιστεύω ναι, μπορούμε να περιμένουμε μια διαφορετική οπτική γωνία από πλευράς των δύο θεσμών. Όταν είναι γνωστές οι συνέπειες της όλης προβληματικής. Μπορείτε να μας πείτε κάτι για την κατάσταση του ιδιωτικού χρέους στην Ευρώπη. Μετά την κρίση έχουν επιδεινωθεί τα πράγματα ή αντίθετα βελτιωθεί λόγω της σταθεροποίησης του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αντολίν. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτή την πρώτη ευκαιρία που έχουμε Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Τρισέ και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο του. Και μια που είμαστε στην αρχή, το μόνο που θα είχα να του ζητήσω είναι να φροντίσει να υπάρχει συνοχή, αλλά συγχρόνως να δώσει και μια νέα θεσμική διάσταση. Οπότε ρωτάω, θα μπορέσετε να τα καταφέρετε. Εμείς θέλουμε και φιλοδοξία και κάθε φορά που βρίσκεται κάποιο κίνδυνο και όταν χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια να μπορείτε να το πείτε. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε μια πολύ σημαντική στιγμή στην ε, ζωή μας. Οπότε θα έπρεπε η φωνή σας να ακούγεται όσο γίνεται πιο γρήγορα όταν πρέπει. Πότε θα είναι η πρώτη φορά που θα μπορέσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Ε, Ευχαριστώ. Και εγώ σας συγχαίρω κύριε Τρισέ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο αυτό το πρώτο σας ε, καθήκον υπό την ιδιότητα του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν η σταθερότητα των ε, τιμών και των νομισματικών αγορών. Τώρα εξετάζουμε δύο κανονισμούς, όπως ξέρετε. Ο ένας έχει να κάνει με τα χρηματοοικονομικά παράγωγα με τις ανταλλαγές πιστοτικού κινδύνου και οι άλλοι με τις ανοιχτές πωλήσει. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε, εσείς θα αξιολογείτε και το κίνδυνο κάθε φορά που πρόκειται για αντισταθμίσεις. Ευχαριστώ. Uh, Αντολίν, τόσο γρήγορα μιλήσατε που εγώ δεν πρόλαβα να ακούσω το τέλος της ερώτησής σας. Μπορείτε παρακαλώ να επαναλάβετε την ερώτησή σας στο τέλος. Την ερώτηση μόνο στην οποία καταλήξατε. Αντολίν, Σχετικά με την ταχύτητα, μπράβο. Ρωτάω, θα μπορέσετε γρήγορα να προχωρήσετε σε πρώτη σύσταση. Πότε θα γίνει αυτό. Thank you. Thank you very much Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω λοιπόν στις τρεις αυτές ερωτήσεις. Τα προβλήματα που παραμένουν όσον αφορά το δημόσιο χρέος. Ναι, πράγματι, να αποτελούν ένα στοιχείο που έχει συστημικές προεκτάσεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και είναι και κάτι που είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να πω, σε επίπεδο ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών. Είναι ένα πρόβλημα που βλέπω εγώ γενικά για τις προηγμένες οικονομίες. Βλέπουμε δηλαδή δυνητικά να δημιουργείται πρόβλημα στις αναπτυγμένες ε, οικονομίες. Γι' αυτό και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Είναι ένα ανοιχτό θέμα δηλαδή. Από πριν βέβαια, αλλά εξακολουθεί. Γι' αυτό και το κοιτάμε. Όσον αφορά τώρα το ιδιωτικό χρέος στην Ευρώπη. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα φαινόμενο «deliveraging» το οποίο δεν ήταν τόσο τραγικό στην Ευρώπη, ήταν λιγότερο δραματικό στην Ευρώπη από τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά είδαμε μια σημαντική μείωση των outstanding πιστώσεων. Σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές έρευνες, δείχνουν μια σταθερότητα στην Ευρώπη στον ιδιωτικό τομέα, τον μη ε, δημοσιονομικό μείον 0,2% όσον αφορά την εξέλιξη αυτή του ιδιωτικού χρέους. Τα νοικοκυριά, βέβαια, διαπιστώνουν ένα σημαντικό βαθμό αύξησης. Αλλά για τον ε, μη δημοσιονομικό ιδιωτικό τομέα υπάρχει μια σταθερότητα. Όσον αφορά τώρα τις παρατηρήσεις που γίνανε για το ότι πρέπει να έχουμε μια καλή διάγνωση αλλά μια διάγνωση που να γίνεται και γρήγορα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Ευρωβουλευτά. Οι κεντρικές τράπεζες, γενικά μιλώντας, αυτές δηλαδή οι οποίες εδρεύουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, αλλά και όχι μόνο, σε ολόκληρο τον κόσμο, οι κεντρικές τράπεζες χρειάστηκε να προχωρήσουν πολύ γρήγορα σε ανάληψη αποφάσεων. Και αν δεν είχαν αναλάβει αυτές τις αποφάσεις, αν δεν τις είχαν λάβει γρήγορα, τις μη τυποποιημένες, θα υπήρχε μεγάλη δυσκολία για τη συνέχιση της νομισματικής πολιτικής με πάρα πολύ σοβαρές συνέπειες. Συνεπώς, επιβεβαιώνω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όπως είπε και ο κύριος Ευρωβουλευτής, να προχωράμε σε σωστή διάγνωση, αλλά έγκαιρα, γρήγορα. Η Επιτροπή, του Συμβούλου Συστημικού Κινδύνου έχει πάρα πολλά ε, μέρη και το κάθε μέρος έρχεται με τη δικιά του εμπειρία, με τη δικιά του αίσθηση του τι επήγει και το τι όχι. Είμαστε μια ομάδα. Εσείς αυτό ζητήσατε, να είμαστε μια ομάδα η οποία ακριβώς να είναι σε θέση να κρίνει όσο γίνεται πιο σοφά. Σοφά, αλλά εφόσον χρειάζεται γρήγορα. Τώρα θέλω να επιμείνω σε αυτό ακόμα περισσότερο. Ακόμα δεν έχουμε αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσουμε και θα εξετάσουμε φτάσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα πιο σύγχρονα και περίπλοκα μέσα, το αναθέτουμε στις ειδικέ αρχές για την αγορά των χρηματοοικονομικών παραγόγων κτλ. Περιμένουμε πολλά από αυτούς δηλαδή, μέσα στην ομάδα, την ευρύτερη ομάδα. Σε αυτό το στάδιο πάντως δεν μπορώ να σας πω πολύ συγκεκριμένα πότε, με κάτι πιο συγκεκριμένο. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές διαστάσεις των αγορών, ότι πολλαπλασιάζονται 5, 6, 7, 8, 9, 10 σε 10 χρόνια αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Εννοείται ότι πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να καταλαβαίνουμε τις εξελίξεις και τις αλλαγές. Την επόμενη φορά σίγουρα θα έχω να σας πω πολύ περισσότερα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ορισμένε ομάδε δεν μπήκανε. Είμαστε, βασιζόμαστε στον κανόνα τυχόν, οπότε δεν μπόρεσαν ορισμένε ομάδε να υποβάλουν το ερώτημά του. Κρίμα γι' αυτό. Κύριε Τρισέ, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σα ξαναδούμε βέβαια σύντομα, υπό τη μία ιδιότητα υπό την άλλη. Και δεν ξεχνάμε ότι έχετε ακριβώ και τι δύο αυτέ ιδιότητε. Σας ευχαριστούμε πολύ πάντω για τον τρόπο με τον οποίο μα εξηγήσατε τα πράγματα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Αστρίντ Λούλινγκ γιατί πρέπει να πάω με τον κύριο Τρισέ σε συνάντηση με την διάσκεψη των Πρόεδρων. Ευχαριστώ. Sei nicht neidisch, es hängt mit dem Alter zusammen, dass ich hier sitze. Μόνο το προνόμιο της ηλικίας είναι που με έφερε εδώ στην ε, Προεδρία, διότι οι διάφοροι άλλοι αντιπρόεδροι δεν είναι διαθέσιμοι. Θα συνεχίσω, αλλά έχω πρώτα ε, ε, ε τη συλλήψεως του λόγου για διαδικαστικό. Έχει το λόγο, κύριε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω να θέσω υπόψη της Επιτροπής το εξής πρόβλημα. Ζήτησα το λόγο για να κάνω ερώτηση εκ μέρους της Γκουε στην προηγούμενη διαδικασία. Σημειωτέων ότι όλες οι ομάδες έκαναν δύο και τρεις ερωτήσεις και η μόνη που δεν έκανε ερώτηση ήταν η Γκουε. Μου δόθηκαν δύο εξηγήσεις Η μία εξήγηση είναι ότι είχε σταλεί ένα μήνυμα και ζητούσε ποιο θέλει να ρωτήσει. Η δεύτερη εξήγηση που έδωσε η πρόεδρος που απεχώρησε πριν από λίγο είναι ότι ακολουθήθηκε ο κανόνας δεχών. Πείτε μου σας παρακαλώ, τι τελικά από τα δύο έχει γίνει. Μήνυμα που να λέει ποιο θέλει να ρωτήσει εγώ δεν έλαβα. Και δεύτερο, αν ο κανόνας δεχόντα αποκλείει μόνο μία ομάδα να κάνει μια ερώτηση τη στιγμή που υπήρχε ο χρόνος να γίνει μια τέτοια ερώτηση. Σας παρακαλώ πολύ, το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το θεωρώ θέμα αντιδημοκρατικής διαδικασίας και θα ήθελα μια υπεύθυνη απάντηση. Oui, monsieur, euh, Αγαπητέ συνάδελφε, μια απάντηση που θα την έχουμε σκεφτεί όρημα θα σας τη δώσει η Πρόεδρος. Περνάμε τώρα Α, παρακαλώ κύριε Λάγκεν. Νομίζω το αίτημα του συναδέλφου μας είναι δικαιολογημένο. Εγώ όμως έχω κάποιος διακόπτη. Έχω μια άλλη ερώτηση ωστόσο. Είναι βρετανική ώρα αυτή εδώ που βλέπουμε στα ρολόγια. Διότι έχουμε Βρετανίδα πρόεδρο. Γιατί λέει εδώ πέρα 3 και 10. Θα το εξετάσω. Θα το εξετάσω. Για ποιο λόγο μας έχουν επιβάλει Βρετανική ώρα και όχι ώρα Βρυξελών. Εν πάση περιπτώσει, προχωρούμε στο υπαριθμό 4 της ημερησίας διατάξεως. Ε, στα αγγλικά μου τα έχουν γράψει εδώ, θα προσπαθήσω να σας τα πω και εγώ στα αγγλικά. 4-9 αγορά με εισηγητή τον κύριο Φεγιό, έχουμε και τους κοιόδης εισηγητάς εδώ. Πρώτος ο κύριος Φεγιό και μετά οι σκιώδεις. Ε, δεν υπάρχει σκιώδη της Γκουε. Όχι, καλά λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα αποφεληθώ από τη δυνατότητα που μου δίδεται για να μιλήσω σύμφωνα με την ώρα Πορτογαλίας. Και εμείς είμαστε πίσω, όπως και οι Βρετανοί. Όμως νομίζω ότι ο Χωσέ Μανουέλ Μαργάιο είχε ζητήσει να μπορέσει να συντάξει την έκθεση για την ενία αγορά, για τις επιχειρήσεις και ήθελα να παρόν για την παρουσίαση μου αυτή. Προφανώς απουσιάζει και μου ζήτησε να αναφερθώ και στο δικό του θέμα για την ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους για τη δική μου γνωμοδότηση. Ευχαριστώ την γραμματεία για τη βοήθειά της, κυρίως την Τζένιφερ Λόγκ. Την ευχαριστώ θερμά για όλη τη βοήθεια που μου έδωσε. Λοιπόν, όσον αφορά τις, ίδιες, ε, τις δύο εκθέσεις έχουν ίδιο στόχο, δηλαδή να γνωμοδοτήσουμε όσον αφορά το θέμα για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς για όλα όσα σχετίζονται με την ενιαία αγορά, όλα τα ζητήματα που αφορούν την ενιαία αγορά, την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και Υπάρχουν διάφορα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σχετικά με το ζήτημα αυτό. Προφανώς εδώ ασχολούμεθα μόνο με μια γνωμοδότηση. Παρ' όλα αυτά η γνωμοδότηση αυτή ασχολείται με πολύ σημαντικά πολιτικά ζητήματα αυτή την παρούσα στιγμή όσον αφορά τη φορολόγηση Φερρυπίν, όσον αφορά τα ευρωομόλογα και διάφορες τροπολογίες και που υπευλήθησαν όσον αφορά την έκθεση του καθηγητού Μόντι Αυτά είναι σημαντικά θέματα και θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι η έκθεση του κυρίου Μαργάγιο όπως και η δική μου, το δικό μου κείμενο θέλουν να πετύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση των πολιτικών κομμάτων. Πολύ συχνά οι απόψεις είναι διαμετρικά αντίθετες για αυτά τα ζητήματα. Όμως, προσέξτε συνάδελφοι το εξή. Εδώ ασχολούμαστε μόνο με μια γνωμοδότηση. Γνωμοδότηση Επιτροπής μας και κατευλήθησαν προσπάθειες για να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή συνένεση. Είμαι ανοιχτό, μπορώ να έχω διάλογο με συναδέλφους αν αυτό είναι αναγκαίο. Είχα όμως και πολλές άλλες υποχρεώσεις και δεν μπορούσα να συναντήσω πολλούς συναδέλφους πρόσωπο με πρόσωπο για να το κουβεντιάσουμε. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Η γνωμοδότηση αυτή πιστεύω ότι μας επιτρέπει να πετύχουμε μια ευρεία συνένεση. Μπορούμε να εθετήσουμε μια θέση που να μας επιτρέψει να συσχετίσουμε τις δύο γνωμοδοτήσεις και θα μπορέσουμε να υποβάλουμε σχετικό κείμενο στην ΙΜΚΟ που θα αντικατοπτρίζει επακριβώς την άποψη της πλειοψηφίας σχετικά με την ε, γνώμη της Επιτροπής μας. Εγώ είμαι έτοιμος να ακούσω ποιες είναι οι απόψεις σας, είμαι ανεκτός Μπορώ να διαβιβάσω τις απόψεις επίσης στον συνάδελφό μας, τον Χωσέ Μανουέλ Γκαρσία Μαργάιο. Η γνωμοδότησή του ακολουθεί παρόμοιες γραμμές όπως η δική μου και μπορώ να του διαβιβάσω τις δικές σας απόψεις. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Ασχοληθήκατε και με τα δύο θέματα από κοινού. Οπότε έχω ένα προβληματάκι όσον αφορά τους κοιόδης συγγητές που είναι οι ίδιοι για την Άντε τους Πρασίνους και την ECR, αλλά όχι για τους σοσιαλιστές θα δώσω το λόγο στο Λίαμ, κύριο Λίαμ Βουανκόκ για την ε, έκθεση Γκαρ, Γκαρσία Μαργάιο και, και ο κύριος Σαμπέν Χουτάς είναι ακολουθή μετά. Λοιπόν, με αυτή τη σειρά θα αναφερθείτε στα δύο κείμενα και μετά η κυρία Γκουλάχ. Σας ευχαριστώ αγαπητή Αστρίτ. Κύριε Ισηγητά, για την γνωμοδότηση αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Φέιο που δούλεψε τόσο γρήγορα και ήδη την προηγούμενη εβδομάδα είχε προτάσεις ε, συμβιβαστικές. Για να πετύχουμε προσέγγιση απόψεων για το θέμα αυτό είναι δύσκολο, οπότε οι προσπάθειές του πράγματι ήταν πολύ καλές. Παρ' όλα αυτά μένει πολλής δρόμος ακόμα για να καταλήξουμε σε συμφωνία που ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Ένα από τα πιο ευαίσθητα πεδία στο θέμα αυτό είναι σίγουρα εκείνο της φορολογίας. Εννοείται ότι πρέπει να απλοποιηθούν τα φορολογικά ζητήματα για τις επιχειρήσεις που δρούν στην εσωτερική μας αγορά. Όμως η κύρια στρέβλωση ανταγωνισμού έρχεται από την απουσία φορολογικής εναρμόνισης και γι' αυτό και στην τροπολογία αριθμό 26 που προτείνω εγώ, προτείνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση όσο γίνεται πιο γρήγορα υπέρ μιας εναρμόνισης των φορολογικών κανόνων. Είναι πολύ βασικό αυτό για την ανταγωνιστικότητά μας. Θέλω επίσης να αναφερθώ εδώ και στην τροπολογία 29 τη Σιλβί Γκουλάρ για τα ευρωομόλογα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή, πολύ σωστή τη σήμερον ημέρα μάλιστα για να ανταποκριθούμε στις κερδοσκοπικές επιθέσεις που δεχόμαστε, όλοι το γνωρίζουν. Τα ευρωμόλογα αυτά όμως μας επιτρέπουν συγχρόνως να χρηματοδοτήσουμε και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020, κάτι που δεν αναφέρεται συχνά. Θέλω να επιστήσω επίση την προσοχή σα στο θέμα τη αλληλεξάρτηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων ε, για τις οποίες δρούν υπεργολαβικά. Είναι πολύ σημαντικέ οι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ιστό, αλλά προσοχή όταν υπάρχει εξάρτηση. Πολλέ από αυτέ βρίσκονται σε σχέση εξάρτηση. Τα διοικητικά θέματα δεν αποτελούν το μόνο εμπόδιο για την ανάπτυξη και την ενίσχυσή του. Πρέπει γι' αυτό να συνειδητοποιήσουμε τις δυσκολίες που δημιουργεί αυτή η σχέση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να φροντίσουμε να έχουμε μια φιλόδοξη πολιτική ώστε να μπορούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να διατηρηθούν στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς και να αναπτυχθούν και όχι μόνο μέσα στην εσωτερική αγορά αλλά και εκτός αυτής. Εξού και η τροπολογία μου αριθμός 21. Και ευχαρίστως να δεχτώ μια αντίστοιχη συμβαστική τροπολογία που περιλαμβάνει το πνεύμα της τροπολογίας μου αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαργάγιο Μαρφίλ για την ε, γνωμοδότησή του. Νομίζω ότι όλα όσα αναφέρει είναι σημαντικά και ενδιαφέροντα. Με απασχολεί όμως το σημείο 4, διότι οι κρατικές ε, επιχορηγήσεις μπορεί να δημιουργήσουν στρεβλώσεις μεν, αλλά όταν είμαστε σε μια κρίση χρειάζονται έκτακτα μέτρα και για ορισμένες χώρες ε, πρέπει να υπάρξουν ειδικά μέτρα. Αυτό για την ε, παράγραφο αριθμός 4 της πρότασης Μαργάγιο Μαρφίλ. Έπειτα κάποια άλλα σημεία θα έπρεπε να συμπεριληφθούν. Η κοινωνική ρήτρα, για παράδειγμα. Ο Μάριο Μόντι μιλάει για την απαραίτητη ε, συμφιλίωση με την κοινωνική διάσταση. Πώς δηλαδή θα επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Γιατί έτσι θα λειτουργήσει η εσωτερική αγορά. Χρειάζεται λοιπόν μια οριζόντια ρήτρα που να περιλαμβάνεται σε όλη την νομοθεσία μας που έχει να κάνει με την ενιαία αγορά άρθρο 9 της συνθήκης εξάλλου, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να οργανώσουμε καλύτερα την αγορά αυτή. Και για να εφαρμόζεται αποτελεσματικά μια τέτοια κοινωνική ρήτρα χρειάζεται μια μελέτη αντικτύπου. Πρέπει να μελετήσουμε όλη την νομοθεσία που έχει να κάνει με την ενή αγορά. Έπειτα χρειαζόμαστε και άλλα μέτρα όσον αφορά την ε, εταιρική διακυβέρνηση. Χρειαζόμαστε στερές εγγύησεις για συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις. Συνεπώς πρέπει να βελτιώσουμε και τις δυνατότητες διαβούλευσης με τους εργαζόμενους. Κάτι άλλο. Όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δουλεύουν μέσα στην ενία αγορά και που θα έπρεπε να αποφεληθούν από πιο ευκολή και καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια θα έπρεπε να μπορούν να υποφεληθούν και από, δημο... και από φορολογικά μέτρα που διευκολύνουν το δανεισμό αυτό. Έπειτα για τις κοινοφελείς υπηρεσίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει πρόταση για να καταγραφούν αυτού του είδου τα μέσα τα οποία θα είναι στη διάθεση των τοπικών αρχών. Τέλος, η γνωμοδότηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και μία πρόταση για καλύτερη προστασία του καταναλωτή. Συγχρόνως βέβαια να προστατεύουμε και τόσες σχήνουν για τον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Κύριε Γκουλάρ για τις δύο εκθέσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς ευχαριστώ ε, διόγκο και στον Χωσέ Μανουέλ θα διαβιβάσω τις ευχαριστίες μου εάν χρειάζονται τροπολογίε, ε, δεν ξέρω αν έχει νόημα όταν θέλουμε να γνωμοδοτήσουμε απλώ, για να μην περιπλέκουμε τα πράγματα. Τώρα, σε σχέση με την ακρόση του κυρίου Τεσέ, θέλω να πω κάτι. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι ζήτησε από τον Ζάκ Τελαροζιέρ και ομάδα εμπειρογνωμόνων να ετοιμάσουν την νομοθεσία όσον αφορά την εποπτεία, κερδίσαμε πολύ χρόνο και καλύφθη πολύ έδαφο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε το ίδιο ζητώντα από τον Μάριο Μόντι, που αυτή τη φορά εργάστηκε μόνο του, και νομίζω ότι υπήρχε μέρημνα για ισορροπία. Ισορροπία μεταξύ διαφορετικών διεκδικήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτών. Να επιτευχθεί ισορροπία. Ο λόγος για τον οποίο η ομάδα μας είναι υπέρ του να ξαναρχίσουμε αυτή τη δουλειά, όχι για να ξαναρχίσουμε το μηδέν, αλλά να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε τα όσα προετοιμάστηκαν από τις εργασίες αυτές τις ποιοτικέ που έγιναν. Εγώ έχω μια ανησυχία βλέποντας ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται προσπάθεια ε, να, να υπάρχει κατακαιρματισμό της προσέγγισης και όχι συνολική προσέγγιση. Και αυτό θέλουμε να υποβάλουμε στην τροπολογία, να υπάρχει συνολική προσέγγιση, θεώρηση. Να έχουμε υπόψη την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές και να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του ανταγωνισμού από τη μια και των απαιτήσεων της δημιουργίας Αγορά με τη θετική έννοια του όρου την άλλη. Δηλαδή να προστατεύονται οι κοινοφελείς υπηρεσίες ή να αναλαμβάνονται κάποιες δράσεις όπως τα ευρωμόλογα. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ περιορισμένο το πλαίσιο και νομίζω ότι αν περάσουμε το σωστό συγκεκριμένο μήνυμα θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να εισακουστούμε. Έχοντας αυτό υπόψη, πρέπει να πω ότι υπάρχει δυνατότητα δυναμικό ανάπτυξη και δυναμικό εξέλιξη, αν θέλετε, όσον αφορά τη μεταρρύθμιση τη εσωτερική αγορά, που θα πρέπει να συνάδει με όσα προσπαθούμε να κάνουμε την οικονομική διακυβέρνηση. Αυτή είναι η θετική πτυχή. Να μην δώσουμε την εντύπωση αποκλειστικά ότι τιμωρούμε βάσει του συμφώνου σταθερότητα στι χώρε και μόνο. Θα θέλουμε αυτέ οι εργασίε να κινούνται παράλληλα με το πακέτο για τη διακυβέρνηση. Αλλά δεν μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα χέρια από τα χέρια του Διόγκο σε αυτό το θέμα. Αυτό ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Πασκάλ Κομφέμ που είναι εισηγητής σκιώδης των πρασίνων όσον αφορά τις δύο αυτές εκθέσεις και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ, όπως και η Σιλβή, θα να πω κάποια πράγματα, να υπενθυμίσω δηλαδή τη σημασία του συμβιβασμού μεταξύ μας και να μην αποκλίνουμε πολύ από την αρχική πρωτοβουλία που ανέλαβε η έκθεση Μόντι και από το πνεύμα που έκανε τι εργασίε του ο Μισελ Μπαρνιέ, που συνάθρισε περίπου 50 προτάσει. Νομίζω ότι θα αποφύγουμε μεταξύ μα να ακολουθήσουμε μια λογική πλειοψηφία κατά μειοψηφία, που είναι το αντίθετο του πνεύματο εντό του οποίου ετοιμάστηκε συνετάχθη έκθεση Μόντι. Ε, και είναι εναντίον τη ε, επίτευξη δυναμικών συμβιβασμών. στο πνεύμα της εκθέσεως Μόντι θέλω να αναφερθώ. Έχω, έχει μια φράση που δεν βρίσκω εδώ στην πρόταση τροπολογία της συμβαστικής τροπολογίας που αρχίσατε να κυκλοφορείτε. Μιλάω για τη συμβαστική σε λατινικό, το σημείο 1α αυτή, Εκεί λέτε ότι καλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαναφέρει το πνεύμα τη εκθέσεω Μόντιο, όπου προωθείται η φιλελευθερωποίηση και ο ανταγωνισμό, ώστε να προωθηθεί η κοινωνική και οικονομική σύγκληση και η φορολογική σύγκληση. Δεν νομίζω ότι το πνεύμα τη εκθέσεω Μόντι είναι ότι πρέπει να προωθήσουμε την φιλελευθερωποίηση και τον ανταγωνισμό που έχει σε συνέπεια τη φορολογική και κοινωνική σύγκληση και την οικονομική σύγκληση. Λέει ότι παράλληλα χρειάζεται εμβάθυνση σε κάποιε διαστάσει τη ενιαία αγορά και ταυτόχρονα χρειάζεται διοργάνωση πραγματική ενιαία αγορά και για τα φορολογικά θέματα. Δεν είναι αίτιο ότι ατό. Είναι παράλληλη λογική που ακολουθείται. Και νομίζω ότι η συμβαστική πρόταση ως έχει συνταχθεί στρεβλώνει κάπω ε, το πνεύμα της εκθέσεως Μόντι. Ένα από τα βασικά στοιχεία του τμήματος για τα φορολογικά και εγώ σχετίζω με αυτό που ελιά Είναι η νέα φορολογική βάση των πολυεθνικών. Ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη του προγράμματο εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2012. Είναι ένα θέμα που είχε τεθεί επιτάπητο από το σύμφωνο ανταγωνιστικότητα που προτάθηκε από την ε, Γερμανία και μετά από τη Γαλλία. Νομίζω ότι αυτό ψηφίστηκε επανειλημμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην έκθεση του Χωσέ Μανουέλ αναφέρεται. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και στη δική σας έκθεση, διότι από ό,τι κατάλαβα την κατανομή των καθηκόντων στη δική σας έκθεση περισσότερο παρά του Χωσέ Μανουέλ θα αναφέρεται, είναι θέμα πυλώνων. Και εδώ δεν βλέπω να γράφεται όμως επισήμως κάτι τέτοιο και θα ήταν επιζήμιο να μην αναφέρεται συγκεκριμένα στο παρόν πλαίσιο όπου πραγματικά εμπεριέχεται συγκεκριμένη πρόταση. Τελευταίο σημείο που αφορά τις κοινοφελείς υπηρεσίες. Είναι μια συζήτηση που συνεχίζεται που αφορά λιγότερο την ΕΚΟΝ αλλά περισσότερο την Επιτροπή Συντερικής Αγοράς που είναι καθήλυνα αρμόδια. Η συνθήκη της Λισαβόνας ενδεχομένως άλλαξε τα δεδομένα όσον αφορά τις κοινοφελείς υπηρεσίες. Υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένε που εμφανίζονται στο Single Market Arc, στην πρόταση του Μισελ Μπαρνιέ και νομίζω ότι συμβασμό που μπορούμε να πετύχουμε είναι ο εξή. Εφόσον ζητάμε συγκεκριμένες προτάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορούμε παράλληλα να ζητήσουμε και συγκεκριμένες προτάσεις για τις κοινοφελείς υπηρεσίες Δηλαδή, τα δύο θέματα ταυτόχρονα τα προωθήσουμε. Αν θέλουμε να απλουστεύσουμε κάποιου κανόνε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, μπορούμε να ζητήσουμε μια απλούστευση κανόνων για τι κοινοφελεί υπηρεσίε που παρέχονται στην τεράστια ψηφία των υποθέσεων όσον αφορά τι κοινωνικέ κοινοφελεί υπηρεσίε που είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, παρέχονται από πολύ μικρέ επιχειρήσει. Θα μπορούσαμε αυτά να τα θέσουμε σαν πακέτο, κοινό πακέτο στι διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ κύριε Κομφέν. Ο κύριος Έπινγκ έχει το λόγο που είναι σκιώδης εισηγητής του ECR όσον αφορά την... και τις δύο εκθέσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα περισσότερα σημεία στις δύο αυτές γνωμοδοτήσεις και συγχαίρω και τους δύο συγκητές. Ο αριθμό των τροπολογιών αναφέρεται στις διάφορες αρχές που έχουν να κάνουν με την νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς, όπως είναι οι τέσσερις ε, βασικές ελευθερίες που πολύ συχνά τις ξεχνάμε. Η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών του κεφαλαίου, των υπηρεσιών και των εργαζομένων. Επίσης, η αμοιβή αναγνώριση είναι και αυτή μια πολύ βασική αρχή για να προχωρήσουμε όσον αφορά την νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς. Υπογραμμίζω επίσης την πολιτική ανταγωνισμού στις τροπολογίες μου που δεν αναφέρεται αρκετά στις δύο αυτές νομοδοτήσεις, θα μπορούσε να υπογραμμιστεί περισσότερο, όπως επίσης και η συνεισφορά, η σημαντική συνεισφορά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτές είναι οι τροπολογίες μου. Πιστεύω ότι είναι επικοδομητικές, μια που συμφωνούν με τη γενική γραμμή και θα μπορούσαν οι συγητές να τη συμπεριλάβουν στη γνωμοδότησή τους. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά με τους σκιώδη συζητές. Η κυρία Κράτσα έχει ζητήσει ακόμα το λόγο. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα απλά να αναφερθώ και εγώ σε δυο τρει δύο, ε, ε, που έχω κάνει σχετικά με το θέμα του πώς οι ενισχύσεις που δόθηκαν ε, στο επίπεδο της εθνικής οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των κρίσεων πρέπει να μελετηθεί πόσο ε, είχαν επιπτώσει τον ανταγωνισμό. Και το άλλο θέμα, πώς υπάρχουν ακόμη στρεβλώσεις, ε, υπάρχουν τομείς όπως η ενέργεια, που σε ορισμένες χώρες επιμένει στην αντίθεση στον ανταγωνισμό, είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν ιδιαίτερα, να δούμε γιατί δεν προχωρεί η απελευθέρωση σε συγκεκριμένους τομείς και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα. Ε, νομίζω ότι είναι δύο θέματα τα οποία αποτελούν στρεβλώσεις ή δυνατότητες στρεβλώσεις και γι' αυτό αναφέρθηκα με τροπολογίες μου. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε καθυστερήσει κάπως και θα ζητήσω από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν έχει κάτι να μας πει από τους παρόντες εκπροσώπους. Κυρία μου, έχετε το λόγο. Σε ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε μια φάση στην οποία ακούει απόψεις και σε αυτή τη φάση οι συνεισφορές των διαφόρων επιτροπών της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς είναι πηγές εμπνεύσεως ε, πολυτιμότατες για τις εργασίες μας για την προετοιμασία της οριστικής εκδοχής για, την, ε, ε, για το νομοθέτημα για την νέα αγορά. Και ακούμε όλες τις απόψεις και τις τροπολογίες με μεγάλη προσοχή. Ε, λοιπόν, πάντα άμα εμπνέεται από εμά και μας ακούει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα θέλω να πω κάποια πράγματα. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν, κυρίως με την αναφορά που, στην ανάγκη που υπάρχει για ένα σαφές μήνυμα που πρέπει να αποσταλεί από την Επιτροπή μας όσον αφορά βασικά ζητήματα που μας αφορούν, ζητήματα που άπτονται της εσωτερικής αγοράς. Και όπως σας είπα, θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και μετά από τη συζήτηση αυτή, τη σύντομη συζήτηση, Πιστεύω ακόμα περισσότερο ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία όσον αφορά τα βασικά ζητήματα. Νομίζω ότι είναι δυνατόν να πετύχουμε μια ευρεία συνένεση στην Επιτροπή μας και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε συστάσεις όσον αφορά το πώς θα πρέπει να λειτουργήσουν τα ευρωομόλογα και όσον αφορά τη σχέση μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πολύ συχνά αναλαμβάνουν υπεργολαβία μικρομεσαίε επιχειρήσεις από τι μεγάλες εταιρείε, Θα διαβιβάσω στον κύριο Μαργάγιο όλα τα ερωτήματα τα σχετικά που ετέθησαν. Και επίσης και για τις κοινοφελεί υπηρεσίες και για, την, για τις οριζόντιες κοινωνικές ρήτρες κλπ. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι κανένας από τους συντάκτες δεν θέλει να αλλοιώσει το όραμα ε, της εκθέσεως ε, Μόντι και θα λάβουμε υπόψη όσα προτάθηκαν. σω οι διατυπώσει των συμβαστικών προτάσεων μπορούν να βελτιωθούν. Θα επεξεργαστούμε τι συμβαστικέ προτάσει, ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αντικατοπτρίζουν σωστά την έκθεση του καθηγητού Μόντι. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Έχετε δουλειά μπροστά σα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι προβλέπαμε, εγώ δεν πρόβλεψα το χρονοδιάγραμμα, ψηφοφορία στις 14 Φεβρουαρίου, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα, Ιστρασβούργων. Πολύ κακή πρακτική είναι αυτή να ψηφίζουμε τέτοια έκθεση σημαντική γνωμοδότηση στο Στρασβούργο διότι τη Δευτέρα το βράδυ υπάρχουν πολλές άλλες συνεδριάσεις και δεν γνωρίζω αν θα μπορέσουμε να έχουμε διαρμην... μετάφραση μάλλον των συμβεστικών προτάσεων σε όλες τις γλώσσες. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τηρήσουμε σωστά τη διαδικασία μας με τέτοιο χρονοδιάγραμμα. Ε, ε, έχουμε η Επιτροπή που είναι καθήλυνα αρμόδια θα ψηφίσει και εκείνη στο Στρασβούργο τη Δευτέρα 17 Μαρτίου. Και αυτό είναι κακή πρακτική. Πρέπει να το πω. Νομίζω θα πρέπει να προσπαθήσουμε αυτό να σταματήσει. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνη όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα, αλλά η Προεδρία θα ήθελα να αναφέρω απλώς αυτά που θα συμβούν. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Και πάμε στο επόμενο σημείο, στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης εταιρική διακυβέρνηση στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς η η κυρία Φόξ, η η κυρία, ο κύριος Φόξ, συγγνώμη, ο κύριος Φόξ, ο κύριος Άσλεϊ Φόξ. Σας δίνω το λόγο, έχουμε τους ε, Σκιώδης, Καντράουι, Μπόλς, δεν είναι εδώ, ίσως θα αντικατασταθεί, Πόρτας, Κομφέ και Μπαζέσκου. Κύριε Φόξ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που συμφωνούμε όσον αφορά το πώς πρέπει να προγραμματίζονται οι εργασίες μας και τι πρέπει να γίνεται στις Βρυξέλλες και τι στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους του Σκιώδης που πήραν το, φρόντισαν να στείλουν τροπολογίες αυτή την έκθεση. Υπήρξε μεγάλη συνεργασία, πολλές λογικές τροπολογίες μου προτάθηκαν και ευχαριστώ την κυρία Πασέσκου την κυρία Μπούλς και τον κύριο Αλκαντράουι που είναι εδώ σήμερα. Ο κύριο Κομφέν θα με συγχωρήσει αν πω ότι δεν υπάρχουν πολλέ από του που μπορώ να δεχτώ. Πιθανότατα διότι ακολουθούμε μάλλον διαφορετική άποψη, έχουμε διαφορετική άποψη στον τον καπιταλισμό. Εγώ το θέλω κάτι καλό και εκείνο θέλει να κρυζώσει τον καπιταλισμό. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι έχοντας εξετάσει τις τροπολογίες βλέπω ότι είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία υπέρ του βασικού πνεύματος της εκθέσεώς μου. Δηλαδή, ότι η διαδικασία, η προσέγγιση η συμμορφώσου ή εξηγήσε θα πρέπει να ακολουθηθεί με διάφορους νομικά δεσμευτικούς κανόνες που θα συνοδεύουν διαδικασία και περισσότερη υποπτία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή σε εθνικό επίπεδο ανάλογα με το ποιο επίπεδο είναι το ενδεικνυόμενο. Θα έλεγα ότι κάποιες από τις τροπολογίες που παρελήφθησαν όσον αφορά αυτή την έκθεση παρεκκλίνουν, βγαίνουν εκτός των αρμοδιοτήτων μας και μπαίνουν εντό τη Επιτροπή Τζούρι, των αρμοδιοτήτων τη Τζούρι, τη Νομική Επιτροπή, όπω το θέμα των αμοιβών. Και θα ήθελα να πω στα μέλη ότι έχουμε μόνο αρμοδιότητα επί συγκεκριμένου θέματο αμοιβών όσον αφορά τα χρηματοστατικά ιδρύματα που έχουν λάβει δημόσια χρηματοδότηση και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να περιοριστούμε σε αυτό το θέμα. Συντάσω τώρα συμβαστικέ τροπολογίες, τις οποίες θα διανύμω στους σκιώδει, το ταχύτερο δυνατόν και μετά ελπίζω να καλέσω τους ε, για να συζητήσουμε αυτές τις συμβαστικέ λύσεις και να καταλήξουμε σε μια θέση που θα είναι αποδεκτή, ελπίζω, από τα περισσότερα μέλη. Κυρία Πρόεδρε, η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα διεξαχθεί στις 13 Μαρτίου και περιμένουμε η έκθεση αυτή να υποβληθεί στην Ολομέλεια το μήνα Απρίλιο. Επειδή έχουμε μείνει πίσω, θα σιωπήσω. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Θα δώσω το λόγο, εντάχει το λόγο του Σκιώδης. Καταρχάς, στον κύριο Καντράουι. Συγγνώμη αν έσφαξα το όνομά σας. Εντάξει κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την παρουσίασή του. Τον ευχαριστώ και για τον τρόπο που δούλεψε. Συνεργαστήκαμε προκειμένου να συμφωνήσουμε σε διάφορα πράγματα. Υπάρχουν όμως ακόμα αρκετές τροπολογίες. Νομίζω ότι ήταν προολικά προσεκτικός για κάποια θέματα. Νομίζω επίσης ότι η διαδικασία του συμμορφώσου η εξήγησε είναι καλή, αλλά θα πρέπει να συνοδευτεί από δεσμευτικά μέτρα, τα οποία να είναι απτά. Γιατί έτσι μόνο θα μπορούμε να έχουμε ένα σωστό και δίκαιο σύστημα. Η συζήτηση είναι τώρα πόσο μακριά θα πάμε, πόσο πολύ θα προχωρήσουμε, πόσο φιλόδοξοι θα είμαστε και αυτό φαίνεται από διάφορα σημεία στα οποία διαφωνούμε με τον εισηγητή. Πάντως πολλές πολιτικές ομάδες συμφωνούν για το ότι πρέπει να έχουμε πιο έντονες τροπολογίες. Για τον κίνδυνο τώρα, η ομάδα μου και εγώ έχουμε υποβάλει διάφορες τροπολογίες ώστε να αποσαφιστούν διάφορα ζητήματα. Το θέμα της ετορικής διακυβέρνησης στα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για την Επιτροπή Κινδύνου, για παράδειγμα, που λέμε ότι θα πρέπει ανεξάρτητα και με πυγμή να μπορούν να δουλέψουν. Συγχρόνως βέβαια χρειάζεται και εποπτεία. Εποπτικές αρχές που να μπορούν να προβούν χωρίς πρόβλημα στο έργο τους και να είναι αποτελεσματικές για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συμμετέχουν εκεί ικανοί άνθρωποι, ικανά στελέχη. Αλλά και ο συλλογικό όργανο πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί ικανοποιητικά και να μπορεί να εκτιμάει σωστά τους κινδύνους. Γι' αυτό και χρειάζεται μια εξωτερική αξιολόγηση για να ξέρουμε κατά πόσο λειτουργεί καλά ή όχι. Τέλος, το θέμα των ε, αμοιβών, των πόνους, δεν ξέρω. Ίσως θα έπρεπε να πούμε κάτι παραπάνω από ό,τι αναφέρεται στην αρχική έκθεση, να αναφέρονται κάποιες αρχές για το πώς θα λειτουργεί αυτό το σύστημα. Πιστεύω και η ομάδα μου ότι χρειάζονται επιπλέον ρυθμίσεις ώστε να περιοριστούν οι συμπεριφορές που οδηγούν σε υπερβολική ανάληψη κινδύνου. Ελπίζω, επιθυμώ, να προχωρήσουμε σε συμβιβασμούς. Είναι πολλές οι τροπολογίες και αυτό ακριβώς δείχνει ότι πρέπει να συνεργαστούμε για να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Καντραουή, λέει η Πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη από το ΕΛΚ, αλλά τώρα μόλις μου είπαν ότι ο κύριος Γκοζές θα αντικαταστήσει την κυρία Μπαζέσκου. Δεν το ήξερα. Οπότε σας δίνω το λόγο ευθύ αμέσως κύριε Γκοζές. Γκοζές. Όχι, δεν σκόπευα να την αντικαταστήσω. Είναι αντικατάστατη εξάλλου, κύριε Μπαζέσκου. Απλώ θέλω να κάνω και εγώ μερικέ παρατηρήσει σχετικά με τι τροπολογίε που κατέθεσε το ΕΛΚ. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι πάμε πολύ γρήγορα. Νομίζουμε ότι η ομάδα μας θα ήταν υπέρ των αρχών που αναφέρονται εδώ και κυρίως της αρχής ε, συμμορφώσου εξήγησε. Είμαστε υπέρ μιας ρύθμισης, αλλά η αυτορύθμιση σήμερα δεν αποτελεί ικανοποιητική απάντηση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Το δεύτερο σημείο τώρα όπου δεν συμφωνούμε και δεν έχουμε στροπολογίε Μπαζέσκου, είναι εκεί όπου η επιθυμεί την εισαγωγή των εθνικών αρχών. Εμείς προτιμούμε ευρωπαϊκές αρχές και θέλουμε η βασική ρύθμιση να είναι ευρωπαϊκή και όχι εθνική. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα για να σας πω ότι η επίτευξη συμβιβασμών μπορεί να είναι πιο περίπλοκη από αυτό που επιθυμεί ο εισηγητής. Αλλά θα φροντίσουμε, τίποτα δεν είναι αδύνατον. Συνεπώς, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε τελικά να καταλήξουμε σε ικανοποιητικούς συμβασμούς. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκοζές. Η κυρία Σάρον Πόλς τώρα που είναι εκ μέρου του Άλντε Σκιώδης θα έπαιρνε το λόγο. Δεν είναι εδώ ούτε και αυτή μπορεί να αντικατασταθεί. αντικατάστατη και αυτή. Δεν βλέπω κανέναν άλλον από το Άλντε να την αντικαθιστά. Οπότε περνώ στον κύριο Πασκάλ Κονφέν και αυτός είναι σκιώδης εισηγητής. Παρακαλώ κύριε Κανφά. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα θα συμφωνήσω με τόσο είπε ο συνάδελφο Ελ Καντραούι. Εξάλλου πολλές τροπολογίες από κοινού τις υποβάλαμε εκείνο και εγώ. Επί τη ουσία η μεγάλη διαφορά είναι τι εμπιστοσύνη μπορούν να έχουμε σε αυτή την αρχή του συμμορφώσου ή εξήγησε. Σε καιρούς κρίσης το να αφήσουμε τις αμοιβέ χωρίς κανόνες δεν θα ήταν καλό γιατί στο κάτω-κάτω αυτό ήταν και το κίνητρο που οδήγησε στο πολλοί να αναλαμβάνουν υπερβολικά μεγάλους κινδύνους. Οι συμβαστικές τροπολογίες δεν πρέπει να είναι άσχετες από τις τροπολογίες που εμείς υποβάλαμε. Υπάρχει και κάποια κόκκινη γραμμή που δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει η ομάδα μας. Θέλουμε ρύθμιση ώστε η Επιτροπή Κινδύνου να μπορεί να έχει πραγματικές εξουσίες για να ελέγχει τους κινδύνους που αναλαμβάνονται από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα μέλη επίσης του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ακόμα εξουσία προκειμένου να ελέγχουν τις αποφάσεις που παίρνουν οι γενικοί διευθυντές. Αυτό σημαίνει μεγάλο περιορισμό της ισόρευσης εντολών των διοικητικών στελεχών γιατί στις διάφορες επιχειρήσεις ή και στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς δεν υπάρχει έλεγχος και τελικά η πολιτική αμοιβών έχει να κάνει με το συμφέρον των επιχειρήσεων και όχι με το συμφέρον των πελατών τους ή ακόμα και αυτών που παίρνουν ε, τις αμοιβέ αυτές. Υπάρχουν ε, πάντως τροπολογίες που παλιότερα έχουμε υποστηρίξει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία και θα ήθελα αυτές να συμπεριληφθούν και εδώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Καμφά. Έχω και τον κύριο Πόρτας εδώ από την ΚΟΕ ως και αλλά δεν τον βλέπω. Οπότε προχωράμε γρήγορα, αφού ο Σκιώδης δεν είναι εδώ. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Φόξ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Α, συγγνώμη, ξέχασα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει κάποιο που θέλει να μιλήσει. Συμφωνείτε να μιλήσει πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. Μας ενδιαφέρουν όσοι ιδέες σε αυτή τη φάση. Ολοκληρώνουμε το Impact Assessment για να κάνουμε πρόταση στον Επίτροπό μας και θα προσανατολιστούμε πιθανότατα επί τριών αξώνων ε, διοικητικό Συμβούλιο, καλύτερη διαχείριση των κινδύνων και εποπτεία αποτελεσματικότερη. Θα τα διαβάσουμε όλα αυτά με προσοχή και θα σας κάνουμε προτάσεις που ελπίζουμε να σας ικανοποιήσουν. Σας ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσες ιδέες που θα αποτελέσουν αντικείμενο προτάσεων προς τον κύριο Μπαρνιέ. Σας έχουμε εμπιστοσύνη λοιπόν, θα κάνετε τα δέοντα. Θα γίνει σωστή διαβούλευση με τον κύριο Μπαρνιέ. Ο κύριος Φόξ έχει το λόγο. Κύριε Φόξ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ακούσατε ποικιλία απόψεων, μεγάλη ποικιλία σήμερα το απόγευμα και είναι η πρώτη φορά που είχα τη δυνατότητα να ακούσω τον κύριο Γκοζές και συνομίλησα με τους βοηθούς της Πασέσκου για το θέμα και θα είναι πολύ δύσκολο όπως καταλαβαίνετε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό επί κάθε πτυχής που συζητήθηκε. Όμως είμαι γενναίος κύριε Γκοζές και θα κάνω ό,τι μπορώ. Merci, euh, Σας ευχαριστώ κύριε Φόξ. Ευχαριστώ που είπατε ότι θα καταβάλλετε μεγάλες προσπάθειες. Σας εύχομαι πολύ κουράγιο και σας συλληπούμε από τώρα στις προσπάθειες που θα κάνετε για συμβαστικές τροπολογίες από τις 144 τροπολογίες που ευλήθησαν. Ευχαριστώ. Περάσω στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή το σημείο 7. Ανοιχτές πωλήσει και συμβάσεις ανταλλαγής πιστοτικού κινδύνου. Ο κ. Πασκάλ Κομφά είναι ο συγητή μα, Θα του δώσω το λόγο και μετά και στους σκιώδη εισηγητέ, αν βέβαια παρίστανται. Ναι, πράγματι έχουμε μείνει πίσω 25 λεπτά. Κάποιοι σκιώδεις εισηγητές θα πρέπει να φτάσουν και σε πιο αργά. Ε, Επαφίεμαι στη σοφία σας. Μήπως πρέπει να διακόψουμε, γιατί προχωρήσαν πιο γρήγορα μάλλον. Εκτός αν θέλετε να ξεκινήσει η συζήτηση με έναν μόνο παρόντα στην αίθουσα, δηλαδή γιατί έχει περιπτώσει εμένα. Ο κύριος Φέρμπερ καταφθάνει, λέει κυρία Λούλινγκ. Ο κύριος Γκέμπελς αντικαθίσταται από τον κύριο Σάντσες Ποσέδο. Ο κύριος Όλε Σμιτ απουσιάζει πράγματι. Ο κύριος Καμάλ απουσιάζει. Και ο κύριος Χέντελ της Γκουε απουσιάζει. Εγώ μπορώ να διακόψω για ένα πεντάλεπτο τη συνεδρίαση και μετά θα δούμε αν θα έχουμε αφήξεις. Καταφθάνει, καταφθάνει. Διακόπτουμε για ένα πεντάλεπτο. Δέκα λεπτά. Για δέκα λεπτά διακόπτουμε. Και ζητώ από τις πολιτικές ομάδες, αν έχουν την καλοσύνη, να φροντίσουν οι σκιώδεις συγητές τους να έρθουν. Ευχαριστώ. Διακοπή για ένα δεκάλεπτο. Oui. Euh, chers collègues, euh, malgré le fait... Λοιπόν, λέει η πρόεδρος, η κυρία Λούλινγκ, η μερίσια διάταξη, μην ξεχνάμε ότι είναι πάντα ενδεικτική όσον αφορά τους χρόνους. Παρ' όλα αυτά, εγώ καθυστέρησα για να έρθουν οι σκιώδες εισηγητέ. Δεν ήρθαν όλοι. Θα δώσω πάντως το λόγο στον εισηγητή για να ξεκινήσει, ο κύριος Καμφά και μετά θα ακούσουμε τους σκιώδεις ηγητές. Το θέμα μας είναι οι ανοιχτές πωλήσει και συμβάσεις ανταλλαγής πιστοτικού κινδύνου. Ο κύριος Καμφά, δεν θα μονοπολίσω το λόγο, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι να ακούσω τις παρατηρήσεις των σκιωδών εισηγητών. Θέλω μόνο να σας πω ότι είχαμε μια πρώτη συνάντηση εργασίας μεταξύ μας, πολύ αποτελεσματική και επικοδομητική. Έτσι καταλήξαμε σε ορισμένε συμβιβαστικέ τροπολογίες. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια δεύτερη τέτοια συνάντηση στο Στρασβούργο και θα ψηφίσουμε στις 28 Φεβρουαρίου και όχι στις 14 όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Επιμένω όμως για το ότι η ψηφοφορία στις 28 Φεβρουαρίου πρέπει να μας επιτρέψει να έχουμε καταλήξει πριν από το Κορεπέρ και το Συμβούλιο που πολιτικά θα επικυρώσουν ε, τις αποφάσεις του κοφή του Μαρτίου. Δηλαδή, η αναβολή αυτή δεν πρέπει να αποδυναμώσει τη θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις διοργανικές συζητήσεις που θα έχουμε με το Συμβούλιο. Κατά τα άλλα, καλύτερα να πάρουν το λόγο οι σκιώδες συζητητές. Οι δύο είναι ήδη εδώ, οι άλλοι δύο έρχονται, είναι στο δρόμο, οπότε τους ακούσουμε. Πρόεδρος, καλώς κύριε Πρώτα απ' όλα το λόγο έχει ο κύριος Σάντσες Πρεσέδο, ο οποίος αντικαθιστά τον κύριο Γκέμπελς, ο οποίος ουσιαστικά είναι αντικατάστατος, αλλά τι να κάνουμε. Θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι λοιπόν προσπαθώ εδώ να αντικαταστήσω τον κύριο Γκέμπελς. ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ, ενώ θα ήθελε, αλλά είναι με κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία στο Λίβανο. Ευχαριστεί τον εισηγητή τον κύριο Κανφέν για το εξαίρετο πνεύμα συνεργασίας με το οποίο ετοίμασε την έκθεσή του. Και όντως και ο κύριος Γκέμπελς θέλει να εκφράσει την ικανοποίησή του για τις συνεδρίες της προηγούμενης εβδομάδας. Αναγνωρίζει ότι κάποιες συμβαστικές τροπολογίες που ακόμα συζητιούνται χρειάζονται παρετέρω επεξεργασία Πάντως μου ανέθεσε να επιμείνω σε τρεις πτυχές που εκείνο θεωρεί ότι είναι αρκετά ευαίσθητες. Πρώτα απ' όλα, το πεδίο εφαρμογή. Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να ενισχύει τον ρόλο των εποπτικών αρχών όσον αφορά όλα τα οικονομικά προϊόντα. Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί κανένα προϊόν, είτε πρόκειται για μετοχές, είτε πρόκειται για ε, συμβάσεις συναλλαγής πιστοτικού κινδύνου, οτιδήποτε, θα πρέπει όλα τα οικονομικά προϊόντα να συμπεριλαμβάνονται και swaps κτλ. Είτε πρόκειται για over the counter, είτε πρόκειται για άλλε μορφέ. Αυτή είναι ξεκάθαρη θέση του. Το πεδίο εφαρμογή πρέπει να είναι ευρύ και να συμπεριλαμβάνονται όλα τα προϊόντα. και ο ιδιωτικό τομέα δηλαδή επίσης πρέπει να εμπίπτει στη ρύθμιση αυτή. Δεύτερον, σε σχέση με τη διαφάνεια του συστήματος αγορών. Πιστεύει ότι χρειάζεται μεγάλος βαθμός διαφάνειας και ότι το σύστημα αγορών είναι αναγκαίο. Δεν πρέπει να αποκλείσουμε τίποτα βάσει της σχέσης κέρδους και κόστους πρέπει οι υποπτικές αρχές να μπορούν να φέρουν σε πέρα στα καθήκοντά τους. Το σύστημα λοιπόν αγορών πρέπει να καλύπτει αυτά που είπαμε. Τώρα κάτι άλλο σημαντικό για τους σοσιαλιστές είναι οι ανοιχτές πωλήσει, short sellings. Εδώ πρόκειται ακριβώς για ανοιχτέ πωλήσει. Δεν είναι ότι είμαστε κατά, όχι, γιατί βοηθούν και προσφέρουν ρευστότητα στην αγορά. Μπορούν να αποτελέσουν ένα καλό δίκτυ προειδοποίησης. Όταν όμως υπάρχει ακάλυπτο, τότε η κατάσταση είναι εντελώ διαφορετική από την κανονική. Γι' αυτό θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας τις επιπτώσεις ενός τέτοιου συστήματος πάρα πολύ καλά. Γιατί στην αγορά δεν υπάρχει μόνο η ζήτηση και η προσφορά. Πολλές φορές επηρεάζουν οι οικονομικοί φορείς την κατάσταση των αγορών, τη ζήτηση και την προσφορά. Γι' αυτό τέτοιου είδου δραστηριότητες μπορεί να είναι αντιπαραγωγικέ. Θέλω επίσης εκ μέρου του κύριου Γκέμπελ να σας πω ότι υπάρχει αισιοδοξία και πιστεύουμε ότι με καλό πνεύμα συνεργασίας θα μπορέσουμε να πετύχουμε μια γενική συμφωνία. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, allé faire Μια που πήγε στο Λίβανο για να κάνει την επανάσταση ο κύριος Γκέμπελς, μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε εδώ. Καθιστυχάστε τον και ελπίζω να υποφεληθεί από τη διαμονή του στην ωραία αυτή χώρα. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Λισμίτ. Α, δεν είναι εδώ. Μήπως υπάρχει κάποιος που τον αντικαθιστά από το Άλτε. Όχι. Ο κύριος Καμάλ τότε. Πού είναι εδώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank Και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο προλαλής σας έπαιξε θαυμάσιο ρόλο. Ε, αντικαθιστώντας ε, τον κύριο Γκέμπελς, με τον οποίο διαφωνώ σε πολλά θέματα, αλλά του εύχομαι καλή επιστροφή από το Λίβανο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πασκάλ για την εργασία του που έχει αναλύσει καλά τον κανονισμό και η συνεργασία μαζί του έγινε σε πολύ καλό πνεύμα. Είναι άνθρωπος συνεργάσιμος και νομίζω ότι πραγματικά οι συμβαστικές προτάσεις που έχουμε κάνει θα έχουν πραγματικά συμβαστικό χαρακτήρα Βέβαια δεν θα είμαστε όλοι απόλυτα ικανοποιημένοι με την τελική έκβαση, αλλά θα είναι ένας ε, εύλογος ε, συμβιβασμός ε, από όλες τις πολιτικές ομάδες που ανεμίχθησαν στην προσπάθεια. Θα ήθελα τώρα να έρθω σε ορισμένα θέματα που με απασχολούν κάπως. Για εκεί δηλαδή όπου ακόμα δεν υπάρχει συμβαστική τροπολογία. για την λεγόμενη locate reserve. Θέλω να δούμε πού θα καταλήξουμε ο συμβασμό. Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε προβλήματα που μπορεί να διώξουν από την αγορά μικρές επιχειρήσεις. Και επίσης, σχετικά με ορισμένες από τις διατάξεις για αυτούς που συμμετέχουν στην αγορά, να γίνουν πιο εύκαμπτες. Αυτό που με απασχολεί πάντως είναι του δημόσιου CDS. Όταν μιλεί κανείς με αρμόδιους στην Ευρώπη, ανισχούν πολύ για ενδεχόμενα ακάλυπτα δημόσια CDS. Να δούμε εάν θα μπορέσουμε να το απαγορεύσουμε. σε μια εποχή που οι κυβερνήσεις ανησυχούν από λόγω του κόστους του δημόσιου δανεισμού πώς θα τις αναγκάσουμε να πληρώνουν ακόμα περισσότερο για, το, για την εξυπηρέτηση του χρέους τους αντί να διαθέτουν τους πόρους για την παροχή υπηρεσιών τέτοιων υπηρεσιών που θα θέλαμε να ε, μπορούν να διαθέτουν και πρέπει να κατανοήσουμε για ποιο λόγο οι θεσμικά όργανα, οι άλλοι οργανισμοί χρησιμοποιούν ακάλυπτα CDS συχνά δεν βρίσκουν κάλυψη, δεν βρίσκουν ασφαλιστική κάλυψη για μια επένδυση και όταν το έργο ε, έχει σχέση με τις πολιτικές της κυβερνήσεως μπορούν να έχουν κάλυψη αν και δεν τις ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ε, σχετικό ομόλογο, αλλά υπάρχει ένα συσχετισμός και ε, με τον κίνδυνο να μην αποδώσει η επένδυση. Μίλησα πρόσφατα με οργανισμούς που χωρίσαν δανειοδότηση για να φτιαχτεί ένα μεγάλο ε, κέντρο καταστημάτων. Αλλά μπορεί όμως η κυβέρνηση να μην ε, καλύψει τελικά. Να μην προσφέρει δηλαδή την ασφαλιστική κάλυψη. Ποια θα είναι η συνέπεια εάν δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τους κινδύνους, τους, κινδύνους τους ή τις ε, επενδύσεις τους. Θα έχουμε τότε απαγόρευση. Εμείς βέβαια θέλουμε να περιορίσουμε τις καταχρήσεις. οι καταχρηστικές συμπεριφορές. Αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το θέμα στην σχετική οδηγία κατά των καταχρήσεων στην αγορά. Αν δεν υπάρχει ο συσχετισμός αυτός. Ή τέλος πάντων μπορούμε να αναζητήσουμε τον συσχετισμό με μια κάπως πιο εξειδικευμένη τροπολογία. Αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι υπάρχει κάποια κερδοσκοπική συμπεριφορά, την οποία δεν θεωρούμε ορθή, μπορούμε να εξετάσουμε επιμέρους περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ε, τράπεζες αναπτύξεως ή ομόλογα από οργανισμούς ή κάποια έργα υποδομής, αλλά θα δούμε πώς θα ψηφίσουν οι δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες. Αλλά και οι σοσιαλιστές και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλουν να καταργήσουν το Sovereign CDS. Αλλά διαρωτώ με ποια θα είναι η επίπτωση στην πραγματική οικονομία. Γιατί θα έχουν κάποια πολιτικά ωφέλη, αλλά θα έχουν κάποια ε, φθηνά πολιτικά ωφέλη εάν απαγορεύσουν κάτι. Αλλά ε, το κόστος για την πραγματική οικονομία ποιο θα είναι. Γι' αυτό ζητώ από τους αδέρφους μου να επανεξετάσουν ποια θα είναι η βίωση στην πραγματική οικονομία και να μην αυξήσουμε τον τρόπο αυτό το κόστος του δημοσίου για το χρέος, για την αντιμετώπιση του χρέους δηλαδή. Καλώς ήρθατε κύριε Σμιτ, που είστε σκιώδης ηγητής των φιλελευθέρων για την έκθεση αυτή και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα τις τελευταίες σας φράσεις κύριε Καμάν. Δεν ξέρω αν θα σας υποστηρίξω. Το θέμα βέβαια είναι πολύ περίπλοκο και δεν υπάρχουν απλές λύσεις. Πάντως πιστεύω και αυτή νομίζω είναι η δική μας ευθύνη και ο Πασκάλ το έχει αντιληφθεί αυτό δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτε εάν δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες γιατί αυτό θα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην αγορά οι διαπραγματεύσεις που διεξαγάγαμε διεξήχθησαν μέσα σε πολύ αξιοπρεπή και φιλική, και φιλική ατμόσφαιρα, σε, σε καλή διάθεση. Από τη δική σας οπτική νομίζω κάνατε ό,τι μπορούσατε. Ίσως πιο μακροπρόθεσμα να μπορείτε να επιτύχετε λίγα πράγματα περισσότερα. Και η γραμματεία μας βοήθησε πολύ. Υποστηρίζω ορισμένες από τις ε, τροπολογίες. για παράδειγμα για την ΕΣΜΑ που βρίσκω ότι είναι πολύ καλή και θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε και περισσότερο νομίζω. Εδώ ίσως μπορείτε να το ξανασκεφτείτε εσείς Πασκάλ, να δοθούν δηλαδή περισσότερες εξουσίες στην ΕΣΜΑ από ό,τι στις εθνικές αρχές. Υποστηρίζω και την πρότασή σας σχετικά με, το, με τις προς το κοινό να περιοριστούν γιατί φοβούμαι ότι οι αποκαλύψεις γιατί οι επιμέρους αυτές ε, ε, αποκαλύψεις οδηγούν σε μια αγελία συμπεριφορά στην αγορά. Και σκέφτομαι αν θα υποστηρίξω την ε, πρόταση διαγραφής των marking orders. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δαπανηρό κάτι τέτοιο. Κάποιος θα πει ότι μπορεί να είναι μια επιχείρηση η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιους διαφορές τελών αλλά μακροπρόθεσμα, και το κόστος δεν είναι πρόβλημα, αλλά εάν περιλάβουμε όλα τα στοιχεία κόστος χωρίς να γνωρίζουμε πώς μπορεί να σωρευτεί το κόστος αυτό στο τέλος, αυτό μπορεί και αυτό να προκαλέσει δυσκολίες στην αγορά. Και έχουμε και το κύριο θέμα για το short selling Εγώ άκουσα στη συζήτηση ορισμένοι συνάδελφοί μας είπαν ότι η τράπεζα Lehman Brothers κατέρευσε λόγω του λεγόμενου naked short selling όπου αγοράζει κανείς ε, μετοχές για να τις πουλήσει αμέσως. Νομίζω ότι το πρόβλημα όμως, το βασικό πρόβλημα το βρισκόταν αλλού και μπορεί να προσέφεραν περισσότερες ε, πληροφορίες για το short selling και να βοηθούσαν την αγορά. Ε, ε, εγώ έχω την δυνατότητα να είμαι μέτοχος σε μια τράπεζα στην χώρα μου και αυτή ήταν πολύ θυμωμένη για το γεγονός ότι γινόταν short selling πριν από ένα-δύο χρόνια και αυτό διότι ή τουλάχιστον αυτοί που διεξήγαν το short selling θεωρούσαν ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στη Βαλτική Και αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να καταργηθεί. Τουλάχιστον το Συμβούλιο και ...η Διοικητική Σύμβουλη. Αλλά εγώ νομίζω ότι σε ένα μικρό ποσοστό το σώτ έλεγχη στην αγορά προσφέρει αξία γιατί μετά από λίγους μήνες εμφανίστηκαν τότε όλα αυτά τα προβλήματα και άλλαξαν. και ο Καμάλ μιλούσε για τα CDS και για τα προβλήματα αρεστότητας και τι θα γίνει με τον κίνδυνο κτλ. Και συμφωνώ. Πριν να κλείσουμε το θέμα αυτό, αυτοί που συμφωνούν μαζί σας θα πρέπει να μας προσφέρουν σημαντικά στοιχεία γιατί το βάρος αποδείξεως βαραίνει εσά ότι δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην αγορά δηλαδή και ότι θα είναι εποφελές για την πραγματική οικονομία. Και ότι τα προβλήματα που εμείς φοβούμεθα δεν είναι παραψευδεστήσεις. Διότι νομίζω ότι ορισμένες από αυτές τεχνικές λεπτομέρειες και ομολογώ δεν ξέρω για τους υπολείπους ίσως όλοι να είστε ειδικοί στον τομέα αυτό αλλά εγώ δεν είμαι δεν είμαι ειδικό στο short selling είμαι μέτοχος σε ορισμένες επιχειρήσεις αλλά δεν είμαι ειδικό για να κρίνω τι έγινε στην αγορά ή τι θα γίνει στην αγορά γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να είστε προσεκτικό και να ακούτε αυτούς που ασχολούνται πραγματικά με το θέμα και που λένε ότι ίσως αυτό να προκαλέσει προβλήματα τελικά στην αγορά. Εγώ επικρίθηκα, όπως ε, μου είπαν, διότι ακούω υπερβολικά την αγορά. Εγώ δεν φοβούμαι να πω ότι ακούω την αγορά, γιατί μια κεφαλαία αγορά η οποία λειτουργεί καλά, οι τράπεζες είναι αναγκαίες για την Ευρώπη αλλά κυρίω η κυβέρνησή μου είναι αυτή η οποία συνεισφέρει στη διαμόρφωση των απόψεών μου. Ορισμένοι μου λένε μην ακούτε τι σκανδιναβικέ κυβερνήσεις γιατί δεν είναι ο αμφαλός του κόσμου. Ασφαλώ, έτσι είναι. Αλλά στη χώρα μου αλλά και στις άλλες σκανδιναβικέ χώρες μπορέσαμε και επιβιώσαμε. Επιβιώσαμε τεραστίων προβλημάτων. Και κανένα πρόβλημα δεν είχαμε με το short selling. Αυτή είναι η άποψη της Σουηδικής κυβέρνησης των εποπτικών αρχών και εγώ βέβαια τους ακούω τουλάχιστον μέχρι ότου να μου αποδείξετε εσείς το ενάντιον. Συμφωνώ πάντως ότι θα πρέπει στην ε, Ευρώπη να υπάρχει μια συμπεριφορά, ένα σύστημα κοινό. Γιατί αυτό που έγινε στη Γερμανία, για παράδειγμα, ήταν πολύ άσχημο. Γι' αυτό να έχουμε ένα σύστημα κωδικοποιημένη συμπεριφορά σε όλη την Ευρώπη. Οπότε μπορούμε να συμφωνήσουμε βέβαια πάνω σε ορισμένους συμβασμούς προς την κατεύθυνση αυτή. Και θα τελειώσω λέγοντας και ούτε θα εκπλήξω κανένα να με το πω αυτό. Είμαστε ισχυρή ομάδα στο κέντρο και εάν εξετάσετε πώς πηγαίνουν οι ψηφοφορίες στο Κοινοβουλίο θα δείτε ότι η ομάδα των φιλελευθέρων ε, κατά το 90 με 95% των ψηφοφοριών ε, βρίσκεται με την πλευρά των νικητών. Δεν είναι περίεργο αυτό γιατί είμαστε κεντρό ακόμα, αλλά υπό τις περιστάσεις αυτές θα έλεγα δεν είμαι καν βέβαιος ότι με υποστηρίζει η ομάδα μου ότι βρίσκεται ακριβώς πάνω στη διαγραμμή όπως εγώ όπως αυτή που σας εξηγώ τώρα Ίσως λοιπόν να υπάρξουν κάποιες εκπλήξεις αλλά θα φανεί αυτό στο τέλος Ελπίζω πάντως Πασκάλ να προχωρήσετε λίγο περισσότερο προς την δική μας κατεύθυνση. Και μην το παρακάνετε. Γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Νομίζω το είδατε ως αστεισμό προηγουμένως και αυτό είναι γεγονός ότι η πολιτική δεν θα πρέπει να καταργούν διάφορους μηχανισμούς, γιατί, να τους απαγορεύουν, γιατί μετά θα πρέπει να απαγορεύσουμε κάτι άλλο. Και τελικά θα καταλήξουμε να ιδρύσουμε μια αρχή απαγόρευσης. Και δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστή στάση ναι, αυτή ναι. της Ευρώπης. Αυτά για την ώρα, Πασκάλ, και προσπαθήστε να κινηθείτε λίγο περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Όλε Σμιτ. Σα εύχομαι να είστε εξίσου πιστικό με του συναδέλφου των, ομάδα σα και ο όπως ε, όσοι ήσασταν εδώ. Ε, Είμαι σίγουρη ότι άκουσε ο κύριος Κομφέν δεόντως αυτά που είπατε. Τις ε, σοφότατες συμβουλές σας. Πρέπει πάντα να ακούτε εκείνους που ξέρουν για τι πράγμα μιλούν. Ε, Έχω ένα πρόβλημα. Καταρχάς ο κύριος Τόμας Χάντλ, κύριε Τόμας Χάντλ της ΚΟΕ, ο σκιώδης ηγετής δεν είναι εδώ. Ο σκιώδης ηγετής του ΕΛΚ, ο κύριος Φέρμπερ, δεν κατέφθασε. Όμως από ό,τι κατάλαβα ο κ. Ζαν Γκοζές, ο συντονιστής μας, ο πολυταλαντούχος, θα τον αντικαταστήσει. Δεν είναι αυτό. Έχει το λόγο. Δεν ζητάω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όχι, όχι, δεν αντικαθιστώ κανέναν. Θέλετε να, να αντικαταστήσω κάποιον άλλο και τώρα τον κύριο Φέρμπερ. Δεν είμαι και τρανσεξουαλικός. Ε, ε, δεν είμαι ούτε συγητής ούτε σκιώδης ε, συγητής. Θέλω απλώς να εκφράσω άποψη. Σαν εκπρόσωπο προ ομάδα μου. Ε, ε, και προσωπική μάλλον, εκφράζω την ομάδα μου. Δεν συμφωνώ τον κύριο Λεσμιτ. Δεν θα είμαι φιλελεύθερο λοιπόν. Λοιπόν, άκουσα τι λέγεται. Λέτε ότι θα πρέπει να δοκιμάσετε αυτό που θέλετε να κάνετε στην αγορά. Καλώς. Καλώς γιατί, αν είναι καλό για την πραγματική οικονομία. 25 χρόνια δικηγόρο είμαι στη ζωή μου και απόδειξε κάτι σημαντικό. Γιατί δεν λέμε ποτέ ότι θα πρέπει η αγορά να αποδείξει ότι αυτό που κάνει είναι καλό για την πραγματική οικονομία. Διότι αυτό είναι καλό ερώτημα. Και ίσω δεν θα απαγορεύαμε, θα παίρναμε διατάξεις για να εμποδίσουμε κάτι που θα θεωρούσαμε ότι ε, θα ήταν καλό για την πραγματική οικονομία. Γιατί είναι μαγική λέξη αυτή η αγορά. Και γιατί αντιμετωπίζετε διαφορετικά από ότι ο καταναλωτής, οι βιομηχανίες, οι λομπίστε. Δέκα χρόνια εργάστηκα σε τράπεζα εγώ. Ε, ήμουνα γενικό γραμματέας και διευθυντή, ενό τμήματο σε μια τράπεζα. Βλέπαμε πάντα ότι δεν ήταν γενικού συμφέροντε οι αποφάσει που λαμβάνονταν και δεν ξέραμε αν ευνοεί το μακροπρόθεσμα από μια απόφαση για την επιχείρηση. Ο όμιλος τον οποίο είχα είχε από 20, μέχρι το 2007 ήταν 23 ευρώ η μετοχή. Ε, τώρα έχει πάει στα 2,80 και 3 η μετοχή. Και ήταν και πολύ συνετές ε, ασφαλείς μετοχές ο οικογενειάρχης αγόραζε για την εξοικονόμηση ε, αυτές τις μετοχές για την αποταμίευσή του, γιατί ήταν καλή τοποθέτηση. Είπατε ότι λαμβάνουν κινδύνου οι μέτοχοι. Τότε θεωρείται αμυντική, ήσυχη μετοχή αυτή που ανέφερα πριν. Γιατί δεν δούλεψε όμως. Γιατί κατέληξε έτσι. Για δύο λόγους. Πρώτον, υπήρχε θηγατρική στη ΣΥΠΑ που ήταν σε μια κατηγορία ασφαλίστρια και άρχισε να ξεγελάει τον κόσμο και να κάνει τα δικά της και μετά έχει επιχειρηματικό μοντέλο, business model, ένα σύστημα εντό το οποίο ε, δανείζαμε μακροπρόθεσμα και εισπάταμε βραχυπρόθεσμα. Λοιπόν, λοιπόν ήταν τελικά τα, οι χρεώστε τα πήγαιναν, οι οφειλέτε τα πήγαιναν καλά. Το επιχειρηματικό μοντέλο τα πήγαινε καλά, οι μέτοχοι τα πήγαιναν καλά. Εάν δεν δείξω την προθεσμία σα, τελικά θεωρείτε ότι είσαστε σε αδυναμία, κατά σε δυναμία πληρωμή. Λειτουργήσε καλά το μοντέλο μέχρι όσου αντιστραφεί η κατάσταση. Και γι' αυτό λέω, πρέπει να αποφύγουμε να απαγορεύσουμε αυτό, θα ήταν παράλογο. Εμείς εδώ όμως θα πρέπει να δούμε τι κάνουν οι άλλοι. Αυτό που κάνουν οι άλλοι, οι αγορές, είναι ορθολογικό, αποδεκτό με την έννοια του κινδύνου. Δεν υπάρχει για τη κατάσταση του κινδύνου. Δεν είμαι υπέρ σοβιετική οικονομία. Αλλά τώρα να λέμε ότι κάθε φορά που έχουμε μια ιδέα θα πρέπει να αποδείξουμε ότι είναι η καλύτερη του κόσμου μέχρι τέλου. Και όταν οι άλλοι έχουν κάποια ιδέα, δεν έχουν τίποτα να αποδείξουν κατά πόσο είναι χρήσιμη η ιδέα του, αυτό είναι ανισόρροπο. Χρειάζεται μια ισορροπία. Σε μια οικονομία που λαμβάνεται η ανάγκη του κέρδου, διότι το κέρδο οδηγεί στην ανάπτυξη στο μέλλον, και θα πρέπει να δούμε ξεκάθαρα να μην δημιουργούμε απόλυτη πραγματική οικονομία. Εγώ δεν είμαι κατά των τραπεζών. Και με ενδιαφέρον διαβάζω τις τροπολογίες που προτείνουν. Πρέπει όμως και να είναι και λογική. Ο Πασκάλ κάτι πρέπει να κάνει για να συναθρήσει τις ιδέες, αλλά δεν πρέπει να παραιτηθεί από ρύθμιση ενός τομέα λέγοντας ότι δεν μπορεί να αποδείξει ότι οι κανόνες που προτείνει είναι σίγουρα επιβλαβείς ή δεν είναι σίγουρα επιβλαβείς για τον τομέα ή θα μπορούσαν. Λένε ότι θα μπορούσαν να είναι επιβλαβείς. Εγώ υποστηρίζω ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να αποδείξουν ε, αυτά που προτείνουν. Αυτά και δεν ήμουν σκιώδης εισηγητής. Βλέπω ότι κατέθεσε κάποιος της ΓΚΟΕ ο Τόμας Χέντελ ήταν σκιώδης εισηγητής. Θέλετε να τον αντικαταστήσετε? Σκιώδης εισηγητής είναι ο σκιώδης Χέντελ της Ενωτικής αριστερά Αριστεράς. Θα λάβετε εσείς το λόγο τώρα για λογαριασμό του. Ωραία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ήρθα με καθυστέρηση γιατί ήμουν και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, ζητώ συγγνώμη. Κάπως αυθόρμητα θα εκφράσω λίγες σκέψεις, αλλά τουλάχιστον ήθελα να πω από τη σκοπιά της δικιάς μας ε, πολιτικής ομάδας ότι για μας δύο πράγματα είναι σημαντικά στην έκθεση του Πασκάλ. Αφενός η απαγόρευση αυτού του λεγόμενου naked ναι short selling, την απαγόρευση την υποστηρίζουμε απολύτως και το άλλο είναι οι κερδοσκοπικές κινήσεις σε τρόφιμα και πρώτες ύλες και άλλα γεωργικά προϊόντα και αυτά πρέπει να απαγορευτούν. Ήδη το θέμα αυτό ξανατέθηκε στις ε, γερμανικές εφημερίδες. Φαίνεται ότι πάλι αυξάνονται οι τιμές των τροφίμων κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο βέβαια να υποστηριχθούν από πλειοψηφία στην Ευρωβουλή τέτοιε ιδέε, αλλά βρίσκω ότι προοπτικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν θα έπρεπε να χάσουμε την ευκαιρία αυτή να περιλάβουμε κάποιες σχετικές ρυθμίσεις ε, στην έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Μεταξύ μας έχουμε εδώ και εκπρόσωπο της Κομισιόν, την κυρία Μαρία Τερέζα Χέλγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπει κανείς εδώ ότι είναι πολύ, ε, πολύ σχηδής η συζήτηση εδώ. Ε, όπως γνωρίζετε η πρόταση της Κομισιόν εγκρίθηκε για να καθιερωθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο το σύστημα συντονισμού μαζί με ένα σύστημα εναρμόνισης μέτρων με σημαντικό ρόλο της ΕΣΜΑ, όχι μόνο στον συντονισμό, αλλά και για την λήψη συγκεκριμένων μέτρων σε περίπτωση που ξεπηδήσουν κίνδυνοι στις αγορές. Τα μέτρα που περιλαμβάνει η πρόταση της Κομισιόν είναι και μέτρα που έχουν ε, προβλεφθεί ανάλογα με, τους, με τα όργανα οι σχετικές σκέψεις της Κομισιόν περιλαμβάνονται στις ε, μελέτες επιπτώσεων που ε, ακολουθούν προσαρτώνται την ε, νομοθετική πρόταση όπως έχει συνταχθεί αυτή είναι πράγματι ανάλογη με τους κινδύνους που ε, ενδέχεται να προκαλέσουν στις αγορές ε, οι διάφοροι μηχανισμοί. Και σε ό,τι αφορά τα μέτρα ε, σχετικά με τους κανόνες locate, η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει ένα Locate rule πολύ αυστηρό. Ανάλογα και με το σύστημα που ισχύει σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε να φύγουν από τις αγορές κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία τους. Αυτό για μας είναι σημαντικό. Να υπάρχει δηλαδή ένας μηχανισμός lock and rule ε, στέρεος. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις διατάξεις marking ή flagging για την διαφάνεια Είναι σημαντικές οι προτάσεις αυτές. Γιατί με την εφαρμογή αυτών των διατάξεων δεν θα υπάρχουν μόνο πληροφορίες στις αγορές ενοποιημένες, αλλά οι αρχές θα έχουν και τη δυνατότητα να λαμβάνουν από τα χρηματιστήρια, από τα trading venues, συγκεκριμένες ειδικευμένες λεπτομερείς πληροφορίες εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, εάν χρειαστεί να γίνουν διώξει για λόγους κατάχρησης της αγοράς. Για μας αυτό το flagging, η επισήμανση δηλαδή, είναι ένα συμπλήρωμα των άλλων μέτρων που προβλέπει η πρόταση αυτή τη Κομισιόν. Εξάλλου, σημειώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αυτό το νομοθετικό μέτρο που συνοδεύεται και από μελέτη επιπτώσεων και όπου βρίσκει κανείς όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα ποιοτικά αλλά και εφικτά διότι τα δεδομένα για τις αγορές σήμερα δεν είναι άφθονα, ας το πω έτσι. Η διαφάνεια ε, των αγορών δεν είναι δεδομένη και Θεωρούμε ότι με μέτρα όπως αυτά που προτείνουμε μέσα στα πλαίσια της ε, ε, απόφασης για το short selling θα οδηγήσουν σε βελτίωση της λειτουργίας των αγορών με όλα αυτά τα μέτρα υπέρ της διαφάνειας, τους κανόνες ε, δικτύων ασφαλείας, ώστε να βελτιωθούν οι λειτουργίες των αγορών αυτών, καθώς επίσης και με τις έκτακτες εξουσίες που χορηγούνται στις χώρες μέλη. Έτσι αυτό δεν είναι απλώς μονάχα θέμα ακαιρεότητας της αγοράς, κατά των καταχρήσεων δηλαδή, αλλά και θέμα σταθερότητας των αγορών. Για την διατήρηση της καλής λειτουργίας υπό πάσαν περίσταση των αγορών. Ευχαριστώ. Έχουμε την μεγάλη τύχη να έχουμε και το σκιώδη εισηγητή του μεγαλύτερου κόμματος και θέλω να τον ρωτήσω αν θέλει και αυτός να παρέμβει. Ο κύριος Φέρβερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ή μήπως είστε πρόεδρος λόγω ηλικίας. Δεν θέλω να παραταθεί περισσότερο η συζήτηση. Οι τροπολογίες που, έχουν καταθέσει, που έχει καταθέσει η πολιτική μας ομάδα είναι ξεκάθαρες. Ακούω πολλά από πλευρά των ενδιαφερομένων κλάδων και για τα CDS. Εδώ βέβαια για τα CDS και την ενδεχόμενη αξία που προσθέτουν διαφωνούν οι ειδικοί. Έχουμε και μια σειρά τροπολογιών ε, τις ε, ρυθμίσεις intraday, δηλαδή αυτά τα στοιχεία μπορούν από μη καλυμμένα να περάσουν σε καλυμμένα μέσα σε μία ημέρα. Βέβαια, πρέπει κανείς να σκεφτεί αν ίσως πρέπει να επιβάλλονται και αυστηρότερες κυρώσεις εφόσον γίνεται σαφώς προσπάθεια παραπλάνησης της αγοράς. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά κατά τη γνώμη μου. Και κάτι που εμείς έχουμε υποβάλει ως πολιτική ομάδα, η ΕΣΜΑ να λαμβάνει θέση για τις, για τις τιμές κατοφλίου να υπάρχει δηλαδή μια διαδικασία εφόσον απαιτείται η ΕΣΜΑ να κάνει κάποιες προσαρμογές. Αυτό έχουμε πει εμείς. Βρισκόμαστε σε εντατικές διαπραγματεύσεις με τον κύριο εισηγητή και ελπίζω το αργότερο στο Στρασβούργο να μπορέσει να αποθρώσει λευκός καπνός από τις καμινάδες μας. Μιας και δεν ήμουν παρούσα ε, στη διάρκεια της συζητήσεως, δεν έχω σημειώσει το όνομά μου στον κατάλογο των αγορητών. Πασκάλ, εσεί πάλι. Πολλά θέματα ετέθησαν που προσπαθούμε να τα καλύψουμε με συμβαστικές ε, τροπολογίες. Δεν θα τα επαναλάβω. Είμαστε μέσω της διαδικασίας θα ήθελα να πω στην Άστριν Λούλινγκ που με κάλεσε να συζητήσω με εκείνους που γνωρίζουν το θέμα. Άστριν, με καλούσατε όταν είσαστε εκεί στο, στη θέση του Προέδρου να μιλώ με εκείνους που γνωρίζουν το θέμα μετά την παρέμβαση του Όλε Σμιτ. Αυτό ακριβώς έκανε. Εκείνοι που ξέρουν καλύτερα το θέμα είναι αυτοί που κινούνται στην αγορά, όχι οι λομπίστες απαραίτητα που έρχονται εδώ και μας βλέπουν, που απλώς μεταφέρουν τις θεσμικές θέσει των ασφαλιστικών εταιριών και των τραπεζών. Θέλουμε να είμαστε οικολογοί και να είναι φίλοι μα αυτοί που είναι εντό τη αγοράς και θέλω να πω ότι πραγματικά αν δεν υπάρχουν πληροφορίε επί του θέματο και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επισήμω στην έκθεσή τη δεν βρήκε τίποτα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα και ότι υπάρχουν κάποιοι που ε, κερδοσκόπησαν όσον αφορά το ΣΕΝΤΕΣ και έπαιξαν με τα επιτόκια για να κερδίσουν και από τα ΣΕΝΤΕΣ και από, από τα ομόλογα. Αυτή είναι η πραγματική η πραγματικότητα εκείνων που παίζουν. Μη φοβάσαστε, έχω συλλέξει τις πληροφορίες. Όσον αφορά τα CDS, θα πρέπει να συζητήσουμε, αν θέλετε, επί του θέματος. Από τη στιγμή που δεν απαγορεύουμε προφανώς τα CDS, όταν υπάρχει υποκείμενο ε, αξιόγραφο, όταν ε, γίνεται χρηματοδότηση στο κράτος, υπάρχει αυτό το ομόλογο που εκδίδεται. Κανείς δεν προ... α... πρότεινε να απαγορεύσει να μην υπάρχει ένα εντές για να υπάρχει κάλυψη. Αν χρηματοδοτεί κανείς το δημόσιο χρέος σημαίνει ότι έχει ένα ομόλογο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μιλάμε για εκείνους που χρησιμοποιούν τα ΣΕΝΤΕΣ χωρίς να χρηματοδοτούν το κράτος διότι δεν υπέχουν αυτή την υποχρέωση και δεν καλύπτονται. Δεν έχουν το χρεόγραφο στα χέρια τους. Το θέμα λοιπόν της κρατικής χρηματοδότησης που αφορά την απαγόρευση του Naked CDS αναμειγνύει την όλη προβληματική. Έχουμε μια φαιά ζώνη των, ε, που πρέπει να συζητήσουμε. Όσον αφορά το marking, σημαντικό θέμα. Εγώ εκπλήσωμαι διότι βλέπω τη φιλελεύθερη που είναι υπέρ τη λειτουργία των αγορών, τη τέλεια και τη διαφανού λειτουργία, όταν θέλουν να δημιουργηθούν τα εργαλεία που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια, ξεφνικά είναι κατά. Όταν μιλάμε για κόστος, το μάρκιν ισχύει στις ΗΠΑ, στο Hong Kong επίσης υπάρχει. Αυτό δεν εμπόδισε την ε, επιβίωση της χρηματοπιστωτικού τομέα ούτε στη ΣΥΠΑ ούτε στο Χονγκ Κόνγκ. Εάν έχουμε περίοδο προσαρμογής, το κόστος θα πρέπει να είναι αρκετά εύκολο να καλυφθεί από τις ευρωπαϊκές τράπεζες που εν τέλει ωφελούνται από ένα προνόμιο αντίθετα από τους Ασιάτες ανταγωνιστές τους στο Χονγκ Κόνγκ και τους Αμερικανούς ανταγωνιστές τους στη Νέα Υόρκη όσον αφορά το θέμα του evidence, αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει marking, κανείς δεν γνωρίζει αν είναι short selling ή όχι. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι ενδεχόμενα παιχνίδια της αγοράς έχουν λάβει η χώρα, δεν υπάρχει χνηλασιμότητα και ακριβώς χνηλασιμότητα είναι αυτή που θέλουμε να εισαγάγουμε μέσω του marking και ακριβώς αυτό ήθελε, δεν ήθελε να κάνει όλο ο Σμιτ. Άρα πρέπει να βρούμε μια λύση όσον αφορά την πρόταση. Εγώ λέω να πάρουμε την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τροποποιώντας την το λιγότερο δυνατόν σε αυτά τα θέματα τα βασικά του marking. Ξέρω ότι διεξάγονται συζητήσεις, δεν έχουμε βρει συμβιβασμό ακόμα, αλλά δεν απελπίζομαι καθόλου, θα τα καταφέρουμε τις επόμενες εβδομάδες που έχουμε από τώρα μέχρι την επόμενη συνεδρίασή μας. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη συνεδρίαση. 5η 10 Φεβρουαρίου, αυτή την εβδομάδα με άλλα λόγια, στις 10 η ώρα. Και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να κηρύξουμε τη λήξη της συνεδριάσεως, αλλά να σας πω ότι στις 6 και 30 υπάρχει άλλη συνεδρίαση εδώ όσον αφορά τον κίνδυνο από όσον αφορά συνεργασία για την χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσετε. Ευχαριστώ.